Good day. Good day. Good morning, Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη Έχουμε φτάσει στο σημείο 12 σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πριν Πρέπει να σας ε, ανακοινώσω ότι πρέπει να, εγκρίνει, να εγκρίνεται τη σύσταση ε, των συντονιστών να διοριστεί η κυρία Σαρτζεντίνη ε, η νέα εισηγήτρια για την ε, πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2009 και 2010, γιατί η πρώην εισηγήτριά μας, η Χάιντι Χαουτάλα, έφυγε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έγινε υπουργό στη νέα φινλανδική κυβέρνηση. Οπότε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση. που έγινε χθε ε, στην συνεδρίαση των συντονιστών. Και αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12, το οργανωμένο έγκλημα. Η εισηγήτριά μας είναι η Σόνια Αλφάνο. Ο στόχος της συζήτησή μας είναι να συζητήσουμε τις ετροπολογίες που έχουν κατατεθεί Οι συντονιστές της Επιτροπής μας αποφάσισαν να συνταχθεί μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Ήταν επίσης αντικείμενο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ακροάσεων που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε στις 12 Απριλίου μια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η εισηγήτρια παρουσίασε τότε την ε, έκθεσή της και η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να ακούσει την άποψη και των εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Και όπως γνωρίζετε, υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός ε, τροπολογιών, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε για να ε, μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε με τη διαδικασία της έγκρισης έκθεσης. Αλλά πρώτα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ήδη είπατε η έκθεση παρουσιάστηκε. Δεν θα μακρηγορήσω τονίζοντας ούτε τη σημασία ούτε την πολυπλοκότητα της θεματικής που αντιμετωπίζουμε. Είναι η πρώτη φορά που αυτού του είδους ε, το θέμα ε, συζητιέται στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η ευθύνη μου επίσης είναι πολύ μεγάλη. Από την άλλη υπάρχει η απόλυτη συνειδητοποίηση ότι αυτό το θέμα, ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ιταλικό. Και ευχαριστώ όλους τους βουλευτές και τους και όδης που κατέθεσαν τροπολογίες. Ευχαριστώ διότι με αυτήν τη συνεχή αντιπαράθεση αποφύγαμε αυτή η έκθεση να θεωρείται ιδιαίτερα ιταλικού χαρακτήρα. Αποφύγαμε η έκθεση να αντιμετωπίζει μόνο ιταλικά προβλήματα και προβληματικές. Έχουμε 243 τρεις τροπολογίες, 75 είναι στο σκεπτικό. Μετά έχουμε και άλλες 100 τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι και εμείς δεχτήκαμε καμιά 80, 20 αποσύρθηκαν ή ενσωματώθηκαν στην έκθεση και έχουμε 34 συμβιβαστικές τροπολογίες. Στις συνεδριάσεις με τους και εισηγητές και κυρίως στη συνεδρίαση της περασμένης ε, Πέμπτης καταφέραμε να μειώσουμε τις τροπολογίες και να τις συνθέσουμε. Εμείς θα θέλαμε να τις ε, συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους σκεώδεις εισηγητές που κατέθεσαν τις τροπολογίες. Ευχαριστώ τους βοηθούς μου, την ε, γραμματεία και τις υπηρεσίες της ομάδας των φιλελευθέρων. Θέλω να ολοκληρώσω ορισμένες πλευρές που μας επεσήμαναν οι εμπειρογνώμονες. Εσείς ε, μας δώσατε, αναφέρατε το hearing της 12ης Απριλίου. Εγώ θέλω να θυμίσω και την ακρόαση της 29ης και 30 Μαρτίου που οργάνωσε η Άλντε και ακούσαμε 50 εισαγγελείς οι εισαγγελείς που ερχόταν και από άλλες χώρες, από την Ισπανία ε, και άλλες χώρες. Μιλήσαμε για, τις, ε, για τη ρωσική μαφία, τη γιαπωνέζικη, την Κινέζικη, την γυριανή. Μιλήσαμε για τη συνεχή παρουσία των μαφιών στο βαλκανικό χώρο και αυτό το οποίο τονίστηκε είναι κάτι το οποίο ήδη το γνωρίζουμε. Αλλά κάποιος ο οποίος δεν, εργάζεται εδώ στο Κοινοβούλιο εντυπωσιάστηκε. Η συνεργασία της δικαιοσύνης ε, και της αστυνομίας χρειάζεται για να καταλήξουμε, δηλαδή της ανακριτικής αρχής μιλάμε, χρειάζεται για να καταλήξουμε σε χειροπιαστά αποτελέσματα ήταν παρόντες από την Ιντερπόλ, από την Ευρωπόλ και ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία γιατί έδωσε ιδιαίτερη σημασία και υποστήριξη σε αυτήν την έκθεση. Αλλά ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει ένα όραμα πολύ πιο προχωρημένο από το δικό μας. Η δικαστικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές προσδοκούν από μας μία εργασία συγκεκριμένου τύπου διότι χρειάζονται μέσα για να αντιπαρατεθούν στο οργανωμένο έγκλημα. Θέλουν να μιλάμε όλοι στις 27 χώρες την ίδια γλώσσα και επί τούτου θα ήθελα να σας θυμίσω τι έγινε χθες. Εχθές στην Ιταλία για την σφαγή του Ντουίσμπουργκ καταδικάστηκαν 7 άτομα σε ισόβια δέσμα. Όλο αυτό ήταν καρπός της συνεργασίας της αστυνομίας του Ντουίσμπουργκ και της ΚΑΠΑ στο Ρέτζο Καλάμπρια. Μπορούμε να πούμε κατά συνέπεια ότι ανταπεξήλθαμε σε αυτήν τη σημαντική ευθύνη που μας ανέθεσαν αλλά μπορέσαμε να δώσουμε και νέες εχμές. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περιμένει κάτι καλύτερο από αυτό και το λέω με ιδιαίτερη ειλικρίνεια. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κείμενο διότι συμμετείχαν ιδιαίτερα οι όδης και πολλοί βουλευτές οι οποίοι συνεισέφεραν. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν επικοδομητικά σχόλια σε αυτό το κείμενο για να μπορέσει να συζητηθεί περαιτέρω το κείμενο και να περάσει στην μήνυ ολομέλεια των Βρυξελών. Ευχαριστώ κυρία Αλφάνο. Υπάρχει και ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο, δεν είναι και υποχρεωτικό, αλλά αν θέλετε ευχαριστώ μπορείτε να πάρετε το λόγο πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, του σκιώδη εισηγητέ και όλου όσου συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή είναι συμβατή με τους στόχους μας και τις προτεραιότητές μας που έχουμε θέσει στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης, όπως επίσης και στο πλαίσιο της στρατηγικής μας ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω την έκθεση αυτή και να σας ευχαριστήσω και πάλι. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ο λόγος ε, στους συναδέλφους. Ο συναδέλφος Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που κατέβαλε για να πλουστεύσει το κείμενο, να το κάνει πιο κατανοητό μέσα από τροπολογίες που συντάσσουμε από κοινού και με τη συνεργασία της Γραμματείας και των σκευών εισηγητών. Είναι η πρώτη φορά που συζητάμε με αυτούς τους όρους για το οργανωμένο έγκλημα. Βέβαια παρά το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστους βουλευτές παρόντες σήμερα. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο ήταν ιδιαίτερα σημαντική κατά τη γνώμη μου. η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών, μεταξύ δικαστικών αρχών, η διαδικασία κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων, η καταπολέμηση φαινομένων ανακύκλωσης του χρήματος, άλλες συγκεκριμένες αναφορές ε, για τα, τη διακίνηση ναρκωτικών, νομοθετικά μέτρα χρησιμοποιώντας τη μαφία κατά της μαφίας και όλα αυτά με συγκεκριμένα και σύντομα χρονοδιαγράμματα. Από την Ιταλία ξεκίνησε η μαφία αλλά το οργανωμένο έγκλημα υπάρχει παντού. Οπότε χρειαζόμαστε τα μέσα ούτως για την εκτέλεση των καταδικαστικών πράξεων κατά της μαφίας παντού. Συνεργασία με τρίτες χώρες για να καταπολεμήσουμε άλλα φαινόμενα οργανωμένου εγκλήματος όπως η σωματεμπορία και το εμπόριο ναρκωτικών. Το κείμενο είναι ευέλικτο, είναι ένα κείμενο το οποίο επιτρέπει σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ειδική νομοθεσία να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτό το κείμενο με έναν τρόπο ευέλικτο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι και για τις τροπολογίες για τις οποίες ακόμα συζητάμε θα βρούμε μία λύση κοινού ενδιαφέροντος, ας πούμε συμβιβασμός για τις δημοπρασίες. Η σκληρή, η αυστηρή φυλάκιση δεν είναι ένα μέτρο βίας κατά του κρατούμενου. Δεν είναι βασανιστήρια ή άλλα τέτοια κακά πράγματα. Απλώς μιλάμε για απομόνωση. Κάποιος ο οποίος είναι μαφιόζος δεν χρειάζεται να επικοινωνεί με τον εξωτερικό κόσμο και να συνεχίζει το οργανωμένο του σχέδιο, το εγκληματικό του σχέδιο. Να τον να του αντιταχθούμε με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Ε, επίσης η κατάσχεση των περιουσιών οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό. Αυτό το μέτρο ισχύει στην Ιταλία και στην Ισπανία θα μπορούσε να γενικευθεί και αλλού. Αναφορά στον δημόσιο τομέα όπου η παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος είναι παρούσα όπως χρειάζονται ε, όπως επίσης υπάρχει και διεφθαρμένη ε, διοίκηση, δηλαδή παράλληλα με τους ε, πολύ σωστούς υπαλλήλου οι οποίοι δουλεύουν για το καλό του, της κοινωνίας έχουμε και πολλούς διεφθαρμένους δίπλα. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτείνει η συγγήτρια πρέπει να το προωθήσουμε. Εγώ όταν μιλούσα για ιταλικό μοντέλο μιλούσα στην, αναφερόμουν στην Ιταλική νομοθεσία η οποία βρίσκεται στην πρωτοπορία διότι στην Ιταλία δημιουργήθηκε το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε νομοθεσίες στην Ιταλία που θα έπρεπε να ληφθούν ε, υπόψη ως ε, σημεία αναφοράς. Είμαι πεπισμένος ότι τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης θα είναι ανάλογα με ε, τις προσδοκίες μας η κυρία Μπορσελίνο. Είναι ε, δύσκολο το έργο της ε, συναδέλφου Αλφάνο διότι πρόκειται για ένα αντικείμενο ιδιαίτερα ευρύ και υπήρξε ο κίνδυνος να βασιστούμε ιδιαίτερα στην Ιταλική εμπειρία. Η Ιταλική εμπειρία που σίγουρα πρέπει κανείς να τη λάβει υπόψη του, διότι δυστυχώς ε, η χώρα μου υποφέρει από πάρα πολύ καιρό από αυτό το πρόβλημα και χρειάστηκε να εξοπλιστεί και να βρει μέσα τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν θα πρέπει να δακτυλοδειχτούμε ιδιαίτερα την μαφία, δηλαδή να επιμένουμε ιδιαίτερα στον όρο μαφία. Η μαφία είναι μία μορφή οργανωμένου εγκλήματος αλλά εξελίχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αν οι μαφίες θεωρώντουσαν πρώτα ένα πρόβλημα όχι της Ιταλίας μόνο αλλά κυρίως της Νότιας Ιταλίας, σήμερα όλες αυτές οι μαφίες έχουν επεκταθεί. Και χάρηκα όταν διάβασα την τροπολογία 134 του κυρίου Κίρχοπ, ο οποίος δεν είναι Ιταλός και μιλάει για τη διακλάδωση της μαφίας με άλλα εγκληματικά δίκτυα και ταυτίζει την μαφία με μια προβληματική εγκληματικής δραστηριότητας διότι πρέπει να μιλάμε σήμερα για οργανωμένο έγκλημα και μαφίες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πλέον όχι μόνο της Νότιας Ιταλίας ή της Ιταλίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί από την πρώτη στιγμή οι μαφίες κατάλαβαν τη σημασία της παγκοσμιοποίησης και παγκοσμιοποιήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι άλλοι λεσοντότητες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τόσο δύσκολη και τόσο πολύπλοκη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα μέτρα, τα οποία χρησιμοποιεί η Ιταλία και είναι δοκιμασμένα μέτρα. Η δουλειά της Σόνια Αλφάνο, κυρίως ε, οι συμβιβαστικέ τροπολογίες, κατέστησαν αυτό το κείμενο πολύ πιο ευέλικτο, πολύ πιο κατανοητό, πολύ πιο εφαρμόσιμο. Νομίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Κροτσέτα. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω και με όσα είπε η συγκήτρια και με όσα είπε η κυρία Μπορσελίνο και ο ο κύριος Γιακολίνο για την έκθεση. Εγώ νομίζω ότι το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο βγαίνει από όλα αυτά είναι ένα καλό κείμενο. Όχι γιατί είναι απλώς ένα εξαιρετικό κείμενο, αλλά είναι ε, μία έκθεση που, στην οποία συνεισέφεραν πολλοί βουλευτές. Μερικά πράγματα όμως θέλω να τα πω, γιατί μετά το διαβάζουμε, την διαβάζουμε την έκθεση ε, και Θα έλεγα ότι διαπίστωσα διαβάζοντας ότι υπάρχουν και ορισμένες προκαταλήψεις γύρω από το θέμα. Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Κανένας από εμά δεν σκανδαλίστηκε όταν οι Ηνωμένε Πολιτείες ζήτησαν να διαβιβάζονται τα τραπεζικά στοιχεία των τρομοκρατών. Κανένας δεν σκανδαλίστηκε τα τελευταία χρόνια όταν η Ισπανία ευνόησε μία, έναν ε, ε, ισχυρό αντιτρομοκρατικό νόμο τώρα τα τελευταία χρόνια διότι είχε το πρόβλημα και κατάφερε αυτό το μοντέλο να το ορίσει ως ευρωπαϊκό μοντέλο. Κανένας δεν θεώρησε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την διαβίβαση στοιχείων για να σταματήσουμε την τρομοκρατία. Εμείς σήμερα συχνά πυκνά στην Ευρώπη και στον κόσμο έχουμε μια κινηματογραφική εικόνα της μαφίας. Εμείς έχουμε όλους αυτούς τους νονούς ε, που κάνουν όλα αυτά τα πολυτελή πάρτι και γιορτές. Καλώς, ε, καλά ανθρωπάκια, άνθρωποι με φιλότιμο, κάτι το έθνικ ε, λαογραφικό φαινόμενο το οποίο μας παραπέμπει σε όλα αυτά τα τοπία της Σικυλίας με μουσικές ε, του 800 που θυμίζει τον Γατοπάρδο, ε, που θυμίζει τέλος πάντων φολκλόρ. Κοιτάξτε να δείτε, οι μαφίες ε, κρατάνε την κοκαΐνη σε διεθνές επίπεδο. Είναι μαφία και οργανωμένο έγκλημα, πουλάνε όπλα και συνδιασυνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία. Και η διεθνής τρομοκρατία δίνει τα ναρκωτικά, δίνει την κοκαίνη και οι μαφίες δίνουν τα όπλα και το οργανωμένο έγκλημα. Οι μαφίες και το οργανωμένο έγκλημα οργανώνουν την σωματεμπορία ε, τη διακίνηση ε, ε, παιδιών, γυναικών που τους πετάνε στους δρόμους στην Ευρώπη κορίτσια τα οποία έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου και που τις υποχρεώνουν στην πορνεία. Όλα αυτά είναι εγκλήματα. Τώρα αυτό το μοντέλο είναι κάτι το απομονωμένο. Πώς μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε τα ναρκωτικά από την Κολομβία μέχρι το Βέλγιο ή μέχρι το Άμστερνταμ. Όλα αυτά γίνονται μόνο γιατί έχουμε μία κολομβιανή μαφία η οποία έχει και το παραστρατιωτικό της ε, σύστημα και στρατό διότι το μοντέλο Όστρα δεν είναι μόνο ιταλικό μοντέλο. Στην Λατινική Αμερική είναι πολύ πιο εκτεταμένο. Έχουμε παραστρατιωτικούς, έχουμε μαφιόζους οι οποίοι είναι και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών Πρόκειται για μια κατάσταση ολοκληρωμένης αποσύνθεσης σε διεθνές επίπεδο. Πέρυσι οι Ηνωμένε Πολιτείε συνέλαβαν 180 μαφιόζους στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Εχθές συνελήφθη στις Βρυξέλλες ένας ε, παράνομος ε, σικελός από το Αγκριτζέντο, από την 50 ε, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου κατοικεί, κοντά στο σπίτι μου <laughs> συγγνώμη κατοικεί και είναι από την ίδια επαρχία με τον κύριο Ιακολίνο. Εμένα μου κόψαν εδώ την... Ε, θέλανε να μου κόψουν τους σωματοφύλακες ε, διότι λέγανε μαφία στο Βέλγιο μπα δεν υπάρχει διότι εμένα η μαφία με καταδίκασε σε θάνατο τελικά διαπίστωσαν ότι υπάρχει μαφία και στο Βέλγιο και με, μα μου την κράτησαν Μα θεωρούμε εμείς ηθικό και μέσα από ένα όραμα ηθικό και αλληλέγγυο της δικαιοσύνης να υπάρχουν πολίτες στην Ευρώπη. Διότι εγώ θέλω να μπορώ να το καταλάβω ότι όποιος κατοικεί στην Ολλανδία ή στη Γερμανία να σκέφτεται ότι το εγκληματικό, όλο αυτό το εγκληματικό πολιτικό φαινόμενο δεν τους αφορά όσον αφορά άλλες χώρες και μετά θα δούμε αν κάτι τέτοιο αληθεύει. Αλλά μπορούν αυτές οι χώρες να παραδεχθούν ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες όπως στη δικιά μου την περίπτωση οι οποίοι ήταν μάρτυρες ε, στα δικαστήρια της χώρας τους γιατί έκαναν καταγγελίες και γι' αυτό βρίσκονται στο στόχαστρο της μαφίας και έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και δεν έχουν προστασία, καμία προστασία στη χώρα τους. Αυτό θέλει να πει η έκθεση. Δεν πρόκειται εδώ να λέμε ότι εντάξει η μαφία είναι στη Γερμανία, στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Όχι βέβαια, διότι μετά και η εθνική περηφάνεια τι λέει, ότι εμείς τόσο χάλια σαν τους Ιταλούς είμαστε. Πρόκειται για χώρες με εντελώς διαφορετική παράδοση και ιστορία, αλλά θέλουμε εμείς όμως να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ αυτών των χωρών, όπου αν κάποιος είναι μαφιόζος, είναι μαφιόζος όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στο Βερολίνο και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες διότι εμείς από οικονομικής πλευράς και εμένα θα μου άρεσε πρόεδρε και το λέω εδώ και θέλω το ξαναπώ θα ήθελα να γράψουμε μία έκθεση για την οικονομική μαφία για του, τις διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικής και νομιμής οικονομίας. Διό, και έχουμε πολλές, διότι όταν τα τοξικά απόβλητα της Γερμανίας καταλήγουν στις χωματερές της ναπολετάνικης μαφίας τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε έναν στρεβλό καπιταλισμό ο οποίος βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση με την εγκληματικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να λέμε ότι εντάξει ναι πρόκειται για ένα εκτεταμένο μοντέλο που δεν είναι μόνο η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες. Σύμφωνοι ξέρουμε ότι έχουμε τη Βαλκανική μαφία, τη Ρωσική μαφία κλπ. κλπ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξή το μοντέλο του οργανωμένου εγκλήματος σήμερα. Όπου και αν βρίσκεται παίρνει ως μοντέλο το μοντέλο της Κόζα Νόστρα. Όπου δεν έχουμε μόνο το έγκλημα του κουρ, δηλαδή διακίνηση ηρωίνης, κοκαΐνης ή εμπόριο όπλων. Αλλά ότι το βρώμικο χρήμα που παράγεται από τις παράνομες δραστηριότητες μπαίνει στην νόμιμη οικονομία και μετά υπάρχουν αλληλοδιασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών δραστηριοτήτων και την, της επίσημης οικονομίας μιας χώρας. Αλλά αυτό όμως συμβαίνει μόνο σε χώρες τις οποίες αφορά το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος. Όχι. Αυτό συμβαίνει παντού, διότι το χρήμα το επενδύουν στις πλούσιες χώρες, εκεί όπου η επένδυση καρπίζει. Βλέπουμε λοιπόν εμείς ότι η μαφία παίρνει τα λεφτά, τα κλέβει τα λεφτά από την ε, Νάπολη, από το Παλέρμο, επενδύει όμως αλλού, στην Ρουμανία, στην Ουγγαρία, στο Μιλάνο, πολύ στις ανατολικές χώρες. Αυτό το μέσο νομίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει αφετηρία. Ένα μέσο επαναστατικό, ανατρεπτικό που θα αλλάξει την ιστορία της νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιτρέψτε μου να πω με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι εγώ δεν... Εγώ δεν βλέπω να γίνεται η σωστή εκτίμηση όλων αυτών των στοιχείων και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση έχει ένα προνόμιο ότι δεν προσποιείται ότι η μαφία δεν υπάρχει. Τελευταίο, για το θέμα της αυστηρής φυλάκισης και την αποκατάσταση των φυλακισμένων. Εγώ ήμουνα και καθηγητής ε, προβληματικών παιδιών, ως εθελοντής δηλαδή ε, δίδασκα παιδιά τα οποία είχαν σχέσεις με τη μαφία και είχα ένα μαθητή 18 χρονών που μου είπε ή πεθαμένος ή φυλακή. Όταν μπαίνει κανείς σε μια οργάνωση της μαφίας δεν βγαίνει ποτέ, δεν υπάρχει αποκατάσταση. Μια φορά που μπήκε, άμα βγεις από την οργάνωση, τέρμα, σε καθαρίζουνε με βάρβαρο τρόπο. Γι' αυτό υπάρχει ο νόμος για τους ε, συνεργάτες της δικαιοσύνης ε, στην Ιταλία. Για να επιτρέπει ε, μια διαδρομή επανένταξης που ξεκινάει από τη διευκρίνηση για το τι εστί μαφία και για το πώς κανείς συνεργάζεται με το κράτος. Δεν υπάρχει αυστηρή φυλάκιση και του λέμε εντάξει θες να αλλάξεις πες μας ό,τι ξέρεις για το οργανωμένο έγκλημα και συνεργάσουμε το κράτος. Όσον αφορά για τις δημοπρασίες, 10 δευτερόλεπτα και τελείωσα. Είναι παράλογο σήμερα μία μαφιόζικη επιχείρηση να μην παίρνει ε, να μην κερδίζει έναν διαγωνισμό στο Μιλάνο, ε, στο Παλέρμο, δεν ξέρω τι, γιατί υπάρχει ο σχετικός νόμος, αλλά μπορεί να κερδίζει έναν διαγωνισμό στο Παρίσι ή στο Βερολίνο ή οπουδήποτε. Λοιπόν, οι μαφιόζοι μας κερδίζουν τους διαγωνισμούς και τις δημοπρασίες σε όλη την Ευρώπη χωρίς κανένας να τους ενοχλεί. Γνωρίζουμε ότι αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντικές για μας, αλλά κυρίως για ορισμένους Ιταλούς συναδέλφους Γι' αυτό είμαστε και ιδιαίτερα γενναιόδοροι στη διαχείριση του χρόνου, κύριε Κροτσέτα. Ο κύριος Άλβρεχτ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω φυσικά την εισηγήτρια να την ευχαριστήσω για την πρότασή της. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα και η καταπολέμηση του οργανωμένου έγκληματος έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και έχει υψηλή προτεραιότητα. Με το θέμα αυτό πρέπει σε βάθος να ασχοληθούμε και ίσως στις προτεραιότητες να καταστήσουμε σαφές ε, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αυτό που είπε ο κ. Κοτσέτα για το οικονομικό έγκλημα το συμμερίζομαι απόλυτα. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να δράσουμε άμεσα με σαφήνεια, με κάθε τρόπο θέλω να πω ότι φυσικά υπάρχει διαφορά εδώ. Αν, στην έκθεση, αν συντάσσουμε έκθεση για την καταπολέμηση της μαφίας ή έκθεση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αν έχουμε έκθεση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να την κάνουμε σωστά με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται οι αρχές μας σε όλα τα είδη του οργανωμένου εγκλήματος και να ταιριάζουν όλα αυτά στο πλαίσιο που συνήθως μέσα στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας και της ποινική δικονομίας όσα ισχύουν. Και φυσικά μια ιδέα σε όλα αυτά είναι, για παράδειγμα, αυτή την υποεπιτροπή ή την ειδική αυτή επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα να θεσπίσουμε, να συγκροτήσουμε. Έχω δυσκολίες όμως αυτή την ιδέα να την βρω απόλυτα σωστή. Όμως, ωστόσο, από την άλλη πλευρά είναι ελκυστική η ιδέα να ασχοληθούμε σε βάθος με αυτό το θέμα. Εξαρτάται από το πώς θα διαμορφώσουμε αυτά τα πλαίσια και αυτά τα πράγματα. Ας αναμείνουμε πρώτα να δίνουμε ποια θα είναι η αξιολόγηση της απόφασης πλαισίου για το οργανωμένο έγκλημα και μετά να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα αιτήματα ή απαιτήσει που θα απορρέουν από αυτό. Με αυτό σίγουρα νέες προοπτικές θα έχουμε που θα απορρέουν και έτσι, από πλευράς πρασίνων, θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε για μια τέτοια δράση. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω για τις συμβαστικές τροπολογίες και για κάποιες από τις δικές μου τροπολογίες. Ιδιαίτερα στο εδάφιο στην παράγραφο 4 και για την απόφαση πλαίσιο για το οργανωμένο έγκλημα εδάφιο 7 και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο 15. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επικρίσεις για αυτή την έκθεση και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο προτού εγκρίνουμε. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τέτοια μέτρα που όπως για παράδειγμα <clears throat> το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερευνών. Εδώ μεταξύ άλλων η ταπεινότητά μου ως σκιώδης εισηγητής ε, για το ευρωπαϊκό αυτό ένταλμα για την άδεια ερευνών, εδώ υπάρχουν μεγαλύτερες επικρίσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με το, άρθρο, ε, με το εδάφιο 9Γ, 9C, όπως διατυπώνεται ότι αυτό το ένταλμα ερευνών υποστηρίζεται λέει απόλυτα από εμά. Δεν το βλέπω έτσι εγώ απόλυτα και πρέπει να είμαστε πιο συνεκτικοί και με μεγαλύτερη συνάφεια για τις θέσεις μας. Αλλιώς θα έχουμε δυσκολίες. Το επόμενο σημείο φυσικά αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταρμα Σύλληψης. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη λειτουργία αυτών των πραγμάτων. Γι' αυτό δεν είναι εύθετο στην παράγραφο 18α, για παράδειγμα, να έχουμε περαιτέρω εξαιρέσεις που προστίθενται που προσθέτουμε περαιτέρω εξαιρέσεις που καταργούμε όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος της αναλογικής χρήσης των μέσων. Όλα αυτά πρέπει με συνεκτικό τρόπο να εφαρμοστούν. Δεν θέλουμε εδώ ένα συγκεκριμένο είδος οργανωμένου εγκλήματος ή την ίδια, το ίδιο το οργανωμένο έγκλημα με περαιτέρω μέτρα να το καταπολεμήσουμε. Αυτό που θέλουμε είναι τα υφιστάμενα μέτρα να τα διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να είναι αποτελεσματικά και να δρουν σωστά και από την άλλη πλευρά να υλοποιούν τις απαιτήσει για το κράτος δικαίου και την ένωμη τάξη. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία όπου είναι σημαντικό να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 2, αυτή η διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος είναι υπερβολικό θα έλεγα αυτό. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε το σφάλμα, να ισοπεδώνουμε τα πράγματα ισοπεδωτικά και να εξομοιώνουμε το ένα με το άλλο συλλήβδιν, έτσι συνολικά το οργανωμένο έγκλημα να το εξισώνουμε με, το, με την τρομοκρατία. Κάπως πρέπει να διαφοροποιούμε περισσότερα τα πράγματα, περισσότερο τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αυτή η έκθεση, ναι μεν, ναι, μεν είναι μια κίνηση για τη συζήτηση, αλλά χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο παραπάνω για να βάλουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε. Διαφορετικά θα έχουμε δυσκολίε και σε άλλε εκθέσει που έχουμε υποσύνταξη. Και θα πρέπει να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ω Επιτροπή δεν το επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κίρκοπ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη που άργησα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ δύο σημεία να θέσω. Το πρώτο είναι το εξής. Μου φαίνεται ότι έχουμε μια συνήθεια να έχουμε όλο και περισσότερες νέες οδηγίες και νέες προσεγγίσεις, ενώ υπάρχουν ήδη ε, δομές ε, στη διάθεσή μας που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε ορισμένα πράγματα. Αν θέλαμε βέβαια να έχουμε ε, καλό έλεγχο και να δείξουμε το σωστό ενδιαφέρον για τις διαδικασίες αυτές. Έχουμε για παράδειγμα σχετική οδηγία από το 2004 που αφορά ειδικότερα το οργανωμένο έγκλημα και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά τη συγκεκριμένη οδηγία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, όταν συζητούμε συνεχώς το ε, οργανωμένο έγκλημα, φοβούμε ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας είναι μάλλον... Ε, ε, βλέπουν κάπως στενόμυαλα το θέμα αυτό και επίσης το βλέπουν στο πλαίσιο των εθνικών τους ορίων. Σε μία συνεδρίαση που είχαμε για το θέμα αυτό, ε, το είχα ξαναπεί, δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιτρέψουμε στην Επιτροπή μας όσο σημαντικά κι αν είναι ε, τα προβλήματα οργανωμένου εγκλήματος σε ένα συγκεκριμένο κράτος, είτε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε είναι η Ιταλία, είτε είναι οι κατοχώρες ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, δεν πρέπει να ε, επιτρέψουμε την εξέβρεση λύσεων για τα συγκεκριμένα προβλήματα μια συγκεκριμένη χώρα. Και αυτό για το οποίο συζητούμε και η Επιτροπή μα είναι πολύ καλή σε αυτό. Συζητούμε για οργανωμένο έγκλημα το οποίο δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα χωρίς να υπάρχει διάκριση από απόψεως ε, ε, των παιδιών που είναι αντικείμενο ε, εμπορίας ε, ε, ή ε, εγκληματικότητας που έχει να κάνει με οικονομικά ζητήματα κλπ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν ευρύτεροι στην προσέγγιση μας. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν θα μπούμε, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα επικεντρωθούμε στην ευρύτερη εικόνα, στη συνολική μας προσέγγιση. Ε, αν έχουμε ήδη ε, κάποια μέσα στη διάθεσή μας, ε, πρέπει ενδεχομένως να διευρυνθεί η προσέγγιση μέσω των συγκεκριμένων αυτών μέσων, να χρησιμοποιήσουμε τις αποφάσεις πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας, πριν ακολουθήσουμε την οδό δημιουργίας νέων. Και ελπίζω ότι είναι η άποψη που θα έχουν και άλλοι συνάδελφοι επί του θέματος. κυρία Αλφάνο για να ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, ξεκινώντας από τον συνάδελφο Γιακολίνο, ο οποίος ανέφερε την οδηγία για τις, ε, για τις δημοπρασίες. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και να βρούμε έναν καλύτερο συμβιβασμό. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία ε, αναφέρει την, την οδηγία για, τις, για τους διαγωνισμούς του 2004 και διαπιστώνω διαβάζοντας την οδηγία ότι κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Διότι εκείνη η οδηγία λέει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Είναι οδηγία του 2004. Αυτή η οδηγία όμως, επιτρέψτε μου αστειευόμενη να πω, ότι εφαρμόστηκε από τα κράτη-μέλη με έναν τρόπο περίεργο είτε με τρόπο χαλαρό είτε με ιδιαίτερα σκληρό ας πούμε σε μερικούς στην, στην Ιταλία σαν την υπόσχεση του, του Καραγκιόζη θα λέγαμε στην Ελλάδα τους ρωτάγανε άμα, α και άμα δεν το ξανακάνεις τότε ορίστε ο διαγωνισμός δικό σου εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πλήρως αυτήν την οδηγία και μέσα σε αυτήν την έκθεση να βρει και ένα σχετικό input. Οι συστάσεις αυτής της τροπολογίας βασίζεται και στα συμπεράσματα της Επιτροπής Ελέγχου ε, Προϋπολογισμού για τη χρήση στα δημόσια έργα του χρήματος του οργανωμένου εγκλήματος. Πιστεύω ότι θα τα βρούμε με τον κύριο Γιακολίνο. Τώρα για την αυστηρή φυλάκιση συμφωνώ με όσα λέει ο κύριος Κίρχοπ. Νομίζω ότι ε, αυτή η τελική εργασία αφορά στο οργανωμένο έγκλημα και τις μαφίες στα κράτη-μέλη και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Απουσίαζε ο κύριος Κύρχοπ και το λέω τώρα ξανά. Η τροπολογία του, η 134, είναι πολύ σημαντική, μιλάει για μαφίες και άλλα διεθνή δίκτυα. Και λέω στον κύριο Άλμπρεχτ, εγώ συχνά ε, αυτά τα χρόνια επισκεπτόμουν Ιταλικές φυλακές και η λεγόμενη σκληρή φυλάκιση, η αυστηρή φυλάκιση, όπως είπαν οι συνάδελφοι, δεν ισοδυναμεί με βασανιστήρια και, αν, και επιτρέψτε μου εδώ οι φυλακές βασανιστήριων είναι ή απλές Ιταλικές ε, ε, φυλακές οι οποίες υποφέρουν από τους υπεράριθμους κρατούμενους. Αυτοί που ε, έχουν αυστηρή φυλάκιση, έχουν μονόκλινα κελιά, έχουν τηλεόραση, εφημερίδες, ε, κλιματισμό και λέμε ότι είναι σκληρή φυλάκιση γιατί δεν έχει επαφές με άλλους κρατούμενους και δεν έχει και επαφές ε, με, με συνδέσμους, με άτομα τα οποία θα μπορούσαν δηλαδή να παίξουν το ρόλο του συνδέσμου με, με τις οικογένειες ε, ή με τις μαφίας ή με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ αν θέλετε θα ανησυχούσα περισσότερο για όλους τους άλλους φυλακισμένους ε, ε, στην Ιταλία οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για χαζά πράγματα με τον νόμο Μπόση Φίνη ας πούμε για το μόνο γεγονός ότι είναι μετανάστες. Και για αυτούς θα ανησυχούσα οι οποίοι δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους, δεν ξέρουν το δικαίωμα ότι μπορούν να έχουν ας πούμε διερμηνία στη δίκη, ότι μπορούν να έχουν μείωση της ποινής και αυτοί εδώ οι φουκαράδες είναι 8 άτομα στις φυλακές, στο κελί. Όταν μιλάμε λοιπόν για αυστηρή φυλάκιση είναι άλλο πράγμα. Και έχει ένα σωρό εκτήματα. Έχει μονόκλινο κελί. Πήγα πριν από 1,5 μήνα σε έναν από τους μπος, σε ένα από τα μεγάλα αφεντικά, τον Τωτόρι Ίνα, ο οποίος μου έδειξε και μου λένε κοίτα, κοίτα να δεις έχω και air condition μου τα ανάψαν κιόλα τώρα αν σκεφτείτε ότι στα Ιταλικά γραφεία, α πούμε, στις δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν air condition, να πούμε στο δικαστήριο του Παλέρμο δουλεύουν χωρίς κλιματισμό, ε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ήθελα να σας το πω αυτό, να έχετε υπόψη σας προστασία των δικαιωμάτων και των μαρτύρων στα δικαστήρια που ανέφεραν η κυρία Μπορσελίνο και Κροτσέτα. Αυτή η εκθεσή εξετάζει την προστασία των δικαιωμάτων και όχι μόνο τα δικαιώματα των οικογενειών, των θυμάτων κλπ. αλλά η προστασία των συνεργατών της δικαιοσύνης, των μαρτύρων. μάρτυρες δηλαδή που είναι αυτοί που καταγγέλουν και οι οποίοι συνεισφέρουν τόσο στο ανακριτικό επίπεδο όσο και στην ε, δικαστική διαδικασία. Και αυτούς δεν τους προστατεύει κανείς ιδιαίτερα. Δεν τους προσέχει κιόλας ιδιαίτερα κανείς. Χαίρομαι που οι πράσινοι και οι ΣΥΕΡ ε, αρχίζουν και ανοίγουν λίγο την ε, αντίληψή τους ε, για την δημιουργία ενός οργανισμού κατά της μαφίας. Και θέλω να τους διασφαλίσω, εμείς δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο όργανο. Ο Άλμπρεχτ πολύ σωστά το είπε Υπάρχουν ένα σωρό οργανισμοί, που είπε και ο κύριος Κύρχο, που ασχολούνται με τα θέματα που ασχολούμαστε κι εμείς. Αλλά αληθεύει ότι αυτοί οι οργανισμοί αναφέρονται στην Eurojust και στην Europol. Δεν έχουν δυστυχώς μεγάλη συνεργασία μεταξύ τους. Εγώ θα ήθελα σήμερα να το τολμήσουμε κάπως. Κάθε φορά που έρχονται εδώ να μας μιλήσουν, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Αυτή ήταν και η αίσθηση που διαμόρφωσα όταν ε, οργάνωσα την ακρόαση του Απριλίου και αυτό επιβεβαίως, μου το επιβεβαίωσε και ένας από τους υπαλλήλους της Ιντερπόλ που ήρθε να μιλήσει αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα προσωρινό νέο όργανο το οποίο θα, θα, θα το ανανεώνει τη φοιτή ανάλογα με τις ανάγκες θα πρέπει αυτό το όργανο να είναι ένα όργανο σύγκρισης αντιπαράθεσης όπως έλεγε και ο κύριος Κίρχοπ να υποστηρίζεται από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Ένα όργανο δηλαδή το οποίο να απαρτίζεται από στελέχη τα οποία θα συντονίζουν όλη την προσπάθεια κατά του οργανωμένο εγκλήματος. Εμείς Προσπαθήσαμε να εντάξουμε όλες τις τροπολογίες. Ε, χθες ο Άλμπρεχτ ε, ανέφερε την παράγραφο 9 ε, γάμα και είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο σκληροί. Εγώ δεν θέλησα να μπω όμως στην ουσία μιας έκθεσης η οποία απλώς προσχεδιάζεται, δεν έχει καθοριστεί ακόμη τελεσίδικα. Γι' αυτό μιλάμε για αντίθεση με το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα, σύγκριση ε, για το να βάζουμε μαζί τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα. Σε αυτήν την τροπολογία εγώ έλαβα υπόψη μου τις σκέψεις άλλων βουλευτών και είμαι πεπισμένη ότι η διασύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας δεν είναι οργανική. Υπάρχει όμως κίνδυνος μία συνέργεια που θα μπορούσε να μας έρθει στο μέλλον, συνεργασίας δηλαδή μεταξύ αυτών των δύο φαινομένων. Γι' αυτό λοιπόν δέχομαι τα συμπεράσματα της ΟΚΤΑ του, ε, ε, του 2011 της Europol. Ευχαριστώ όλους τους και όλες όλους τους συναδέλφους που κατάθεσαν τροπολογίες. Με μία τελευταία αναθεώρηση των παρατηρήσεων, Νομίζω ότι τα είπα όλα. Ναι, ναι. Μου φαίνεται να τα είπα όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να φροντίσουμε το χρόνο, λέει ιταλικά ο πρόεδρος. Βέβαια τώρα ξέρετε και εμείς ε, μετά από αυτά που μας είπατε για τον κλιματισμό του κυρίου Γιακολίνο, ε, του κυρίου Τωτόρι Ίνα, ο, ο κύριος Γιακολίνο θέλει να πει κάτι. Διευκρίνηση σύμφωνοι στην αυστηρή, με την αυστηρή φυλάκιση που οδηγεί στην απόλυτη απομόνωση. για την καταστολή αυτών των μαφιόζικων εγκλημάτων. Τώρα για την ε, κανονική φυλάκιση μπορεί να πει κανείς ότι στην Ιταλία καλύτερα κανείς να είναι μαφιόζος από ότι φυλακή, απλώς φυλακισμένος. Στην Ιταλία από τις πόσες χιλιάδες κρατούμενους το 1 τρίτο προέρχεται από, από τρίτες χώρες. Στις 10-11 Δεκεμβρίου του 2009 προβλέψαμε εδώ στο Κοινοβούλιο με μια τροπολογία κονδύλια για τα κράτη-μέλη για την επέκταση και αναπαλαίωση των φυλακών λόγω της αύξησης των κρατουμένων και κυρίως από τρίτες χώρες. Εγώ μίλησα με την αρμόδια διευθύντρια ε, που ασχολείται με το θέμα και μου είπε ότι με τις νέες προοπτικές του 2014 δεν ήταν ο κλιματισμός, ήταν το θέμα. Μπορεί να φέρεται ως ανέκδοτο δηλαδή, αλλά δεν είναι. Ξέρω ότι ο υπερπληθυσμός στις φυλακές δεν είναι μόνο ένα ιταλικό πρόβλημα. Α, ξέχασα κάτι πριν και το λέω τώρα δηλαδή. Καλό θα ήταν να έρχονται τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μετά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να το ρίσουμε όλα αυτά. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν με τη συζήτηση. Επόμενο σημείο. Για την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση ουσιών που είναι πρόδρομοι εκρηκτικών υλών. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό είναι ο Ιαν Μούλτερ και είμαστε εδώ για να εξετάσουμε την, ε, το σχέδιο γνωμοδότησης σε σχέση με την αγορά και χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρητικών υλών. για τη μείωση της πρόσβασης του Εβραίου κοινού σε υψηλού κινδύνου ουσίες ε, και ειδικότερα για ουσίες ε, που μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά οικιακής κατασκευής. Οπότε ας ακούσουμε τώρα την παρουσίαση της γνωμοδότησης από τον κύριο Μούλτερ και μετά ε, να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ευπρόσδεκτη και επίσης νομίζω ότι καλό είναι το γεγονός ε, ότι είναι κανονισμός και όχι οδηγία, γιατί ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Όταν λοιπόν ε, θα εφαρμόσουμε την πρόταση αυτή θα μειώσει την ε, πιθανότητα ε, τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών με χημικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πραγματικά για αυτό το λόγο είναι πολύ ευπρόσδεκτη πρόταση. Ο κατάλογος των ουσιών που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σχεδόν πλήρη. Εγώ τρει με τέσσερι μήνε ε, περίμενα μήπως ο κλάδος ε, υποβάλει και άλλες προτάσεις, αλλά πρέπει να πω ότι όλοι όσοι ήρθαν στο γραφείο μου μου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με τον κατάλογο των ουσιών, γιατί ήταν σχεδόν πλήρης. Επομένως δεν χρειάστηκε εγώ να ε, καταθέσω πολλές τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, έκανα μία πρόταση να σεβαστούμε πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων από τις αρχές Μαρτίου χρονολογείται για να χρησιμοποιήσουμε την ίδια διατύπωση και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ε, κάθε δυνατότητα να αλλάξει τον κατάλογο των ουσιών και τότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν ε, να διαφωνήσουν ε, εάν θεωρήσουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Συνεπώς, οι τροπολογίες που θα καταθέσω και τις οποίες δεν έχετε ακόμη στη διάθεσή σας, κάποιος μου είπε μάλιστα πώς ακριβώς ορίζεται ε, την ύποπτη συμπεριφορά και βρίσκω λίγο δύσκολο τον ορισμό αυτό να σας πω την αλήθεια και περιμένω κάποιοι συναδέλφους να μου πούν και εκείνη την άποψή τους ε, για να έχω μια καλύτερη, έναν καλύτερο ορισμό του τι είναι ύποπτη συμπεριφορά ώστε κάποιος ε, που βλέπει κάτι σε μια συναλλαγή που δεν τη θεωρεί απολύτως ασφαλή να μπορεί στο εθνικό σημείο επαφής να την καταγγείλει. Αυτά όσον αφορά λοιπόν το, ε, το επίπεδο κινδύνου των ουσιών θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν ε, την προστασία του ιδιωτικού βίου των ε, ενδιαφερομένων. Πρόκειται λοιπόν για στοιχεία που θα αφορούν ε, την ασφάλεια των δεδομένων και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών. Προτείνω λοιπόν μία περίοδο δύο ετών για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, εν συντομία τα σχόλιά μου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία πιστεύω, όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι ε, ευπρόσδεκτη και πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μόλντερ. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε και την, τον εκπρόσωπο συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ντίκ Χάιμανς και είναι και εδώ εκπρόσωπος ε, της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Μήπω θέλει κάποιο από το Συμβούλιο να πάρει το λόγο σε αυτή τη φάση. Α, όχι. Εντάξει τότε, να περάσουμε στους συναδέλφους. Κυρία Ματιού, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Θα ήθελα να θέσω τέσσερα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Για ποιο λόγο έχουμε περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ε, στο ευρύ κοινό ε, και δεν, ε, το δεν έχουμε συμπεριλάβει και τους επαγγελματίες, μια και πρόκειται για θέμα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Υπάρχει επίσης και ένα θέμα... Ε, καταγραφή σε ένα συγκεκριμένο μητρό ε, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μία ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα 1. Όμως ε, αναφέρεται το άρθρο, στο άρθρο 3 ότι κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο, οργάνωση ή ένωση ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει νόμιμα μία τέτοιου είδους ουσία αν αυτή δεν απαγορεύεται στον κανονισμό. Είναι πολύ εύκολο όμως να γίνει κάτι τέτοιο σε ορισμένα κράτη-μέλη και γι' αυτό ακριβώς ε, προτείνω στον κανονισμό να, συμπεριληφθεί, ε, να συμπεριληφθούν όχι μόνο τα νομικά και φυσικά πρόσωπα αλλά και οι επαγγελματίες του κλάδου. Ε, επίσης ο κανονικός προβλέπει ότι αναφέρονται στο παράρτημα 1 όταν η συγκέντρωση υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο ε, και όταν υπάρχει αδειοδότηση για τον παραγωγό της ουσίας ε, τριετούς ε, διάρκειας. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου χώρα, τη Γαλλία, το 2009 1.250.000 ιδιωτικές πισίνες υπήρχαν στη Γαλλία και φαντάζομαι ότι στα κράτη -μέλη, σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν εξίσου πολλές πισίνες για τον καθαρισμό των ε, της πισίνας για παράδειγμα ε, χρησιμοποιείται ένα προϊόν το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα 1 δεν είναι ιδιαίτερο οικολογικό το προϊόν αυτό και παρουσιάζει σημαντικά ε, πλεονεκτήματα σε σχέση με το χλώριο τα συμβόλαια των, της συγκεκριμένη άδεια δίνουν διάρκεια χρήσης τους τεράστια για ποιο, για ποιο λόγο λοιπόν να μην δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα πρόληψη και προστασία ε, που θα ήταν πιο ευέλικτο, που θα δίνει στη δυνατότητα στου ε, αγοραστέ των συγκεκριμένων καταγεγραμμένων ουσιών να δηλώνουν την νόμιμη χρήση που θέλουν να κάνουν ε, του συγκεκριμένου προϊόντος. Οπότε οι υποχρεώσει που προβλέπει ο κανονισμό για να υπάρχει ένα μητρό των, πολι... των πωλήσεων των ουσιών αυτών και, και καταγγελία των συγκεκριμένων ύποπτων συναλλαγιών Λοιπόν θα επέτρεπε την ανιχνευσιμότητα των πωλήσεων, αλλά θα έπρεπε αυτό να αφορά όλες τις αγορές και από τους επαγγελματίες και από τους ιδιώτες και όχι μόνο ο ιδιώτης να ε, έχει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Το τρίτο σημείο αφορά το παράρτημα. Η πρόταση κανονισμού που αναφέρει ε, την... Ε, ε, συμπερίληψη στο παράρτημα δύο ε, ουσιών που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη συγκέντρωση και στο παράρτημα 2 αναφέρονται όλες οι ουσίες τις οποίες πρέπει να αναφέρουν οι αγοραστές. Ε, εγώ, εμείς πιστεύουμε ότι δύο διαφορετικές λίστες, δύο διαφορετικοί κατάλογοι δεν έχουν επιστημονική βάση, διότι ο κίνδυνος που αναφέρεται στο παράρτημα 2 ε, δεν είναι διαφορετικές ε, από το παράρτημα 1 από απόψεως επίπεδου συγκέντρωσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα λιγότερο περιοριστικό ε, πλαίσιο και θα ήθελα να αναφερθώ και στο τελευταίο σημείο που με απασχολεί για το άρθρο 6 παράγραφος 4 που λέει ότι πρέπει να αναφέρεται κάθε ύποπτη συναλλαγή των ε, καταγεγραμμένων προϊόντων, τι γίνεται με τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ε, μη βιομηχανικής κατασκευής γιατί ε, πρέπει ο πολιτής να εκτιμήσει κατά πόσο πρέπει να καταγγείλει την ε, χρήση μιας ουσία που δεν αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού. Κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει μη ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού, γιατί είτε αναγνωρίζεται η ουσία από μια συγκεκριμένη συγκέντρωση και πέρα που θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκρηκτικό, για τη, χρήση, για τη δημιουργία εκρητικού, ε, όμως είναι αρκετά χαλαρή αυτή η εφαρμογή γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ε, ενιαία εφαρμογή του κανονισμού ε, όπως αναφέρεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε De έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλντε για το σχέδιο έκθεσης. Και όσον αφορά και τα delegated acts, είναι το γνωστό κείμενο κατ' κατεντολήν πράξεων ή κατεκτέλεση. Τρεις πτυχές πρέπει να δούμε. Προστασία δεδομένων, προστασία ιδιωτικής ζωής ή σφαίρας και έχουμε μια γνωμοδότηση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Μεσολαβητή, Διαμεσολαβητή δεν βρήκε ακόμα την απήχησή του αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα. Πώς το σημείο δηλαδή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τι θα κάνουμε, ποια περίοδο, ποιο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα. Βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, είμαι ένας ας πούμε έμπορος ε, στο λιανικό εμπόριο και θέλουμε να θεσπίσουμε κανόνες ε, και ε, κανονισμούς που θα ισχύουν και για τους ε, εμπόρους στο λιανικό εμπόριο και όχι μόνο για τους μεγάλους, ε, για τους εμπόρους Θα πρέπει να εξετάσουμε να δούμε είναι κάτι ύποπτο ή τι γίνεται. Θα πρέπει ουσιαστικά καθημερινά να γίνεται αυτό με κάθε πολίτη. Έτσι δεν είναι. Γιατί διαφορετικά δεν θα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες. Πρέπει να βλέπουμε, είναι σεβαστοί από όλου οι κανόνες ή όχι. Δηλαδή, να δούμε, είναι βιώσιμος ο κανονισμός αυτός, είναι εφαρμόσιμος. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφής ο κανονισμός και οι διατάξεις του. Και δεν, είμαι, δεν έχω τη βεβαιότητα ότι συμβαίνει αυτό θα έπρεπε να δούμε και τις οργανώσεις των ε, καταναλωτών και να τις ακούσουμε. Για παράδειγμα, στον κατάλογο βρίσκεται και το ασετόν. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται συχνά, δεν είναι τίποτα ύποπτο αν πουλάει κανείς ασετόν. Όμως παρόλα αυτά μπορεί να είναι κάτι το επικίνδυνο αν χρησιμοποιηθεί ε, με, με κακό τρόπο, με επικίνδυνο τρόπο. Πρέπει λοιπόν την εφαρμοσιμότητα, την υλοποίηση και το εφικτόλων αυτών να το εξετάσουμε σε βάθος, να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν και τώρα έχετε τον λόγο εσείς για να απαντήσετε σε αυτές τις παρατηρήσεις, εσείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω μια προκατακτική απάντηση στα θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση. Πρώτο, αυτό της κυρίας Ματίω, το εύρος του κανονισμού. Το θέμα γιατί οι επαγγελματικοί χρήστες αποκλείστηκαν από το εύρος αυτού του κανονισμού. Η απάντηση είναι σχετικά απλή. Συγγνώμη. Λοιπόν, η απάντηση είναι σχετικά απλή. Είχαμε πάνω από δύο χρόνια συζητήσεις με επαΐοντες και πραγματογνώμονες από τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις απειλές από πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών. Και ήταν σαφή αυτά που είπαν ότι οι κύριες απειλίες, απειλές προέρχονται από εκείνους που αγοράζουν αυτά τα χημικά, σε ένα, τις χημικές ουσίες σε ένα μαγαζί και όχι εκείνους που τις χρησιμοποιούν χονδρεμπορικά. Οι ιδιώτες δηλαδή στις αγορές τους χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα και γι' αυτό οι διατάξεις για τις ύποπτες ε, συναλλαγές εφαρμόζονται σε όλες αυτές τις ουσίες και εφαρμόζονται και για τους επαγγελματικούς χρήστες. Υπάρχει ένας συνδυασμός διαφορετικών μέτρων και όταν έχουμε αυτορύθμιση που περαιτέρω θα καθιστούσε πιο ασφαλή αυτή την αλυσίδα συναλλαγών από ό,τι μέχρι σήμερα. Ακολουθώντας αυτές τις ευρύτερες ε, διαβουλεύσεις θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Οι διαφορές μεταξύ αδειών και καταχωρήσεων. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, θα γίνει κατανοητό. Αν ε, υποβάλει αίτηση κάποιος, έχουν οι αρχές ευκαιρία να δουν αν έχει κάποιος ένα ποινικό μητρό βεβαρημένο. Μπορούν να δουν αν υπάρχουν πληροφορίες ε, για κάποιο άτομο που μπορούν να καταστήσουν επικίνδυνο αυτό το άτομο ή να το αποκλείουν ε, για την αγορά τέτοιων ουσιών με ένα τέτοιο σύστημα καταχώρηση, με ένα σύστημα, χωρίς ένα σύστημα καταχώρησης οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει ε, μια τέτοια ουσία ή αν υπάρχει απλώς και μόνο μια ε, καταχώρηση πάλι δεν μπορεί να υπάρξει η ταυτοποίηση και γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει η βεβαίωση ότι αυτά θα γίνονται. Ξέρουμε ότι τα θέματα τα οποία αφορούν τη χρήση αυτών των χημικών ουσιών αφορούν την καθημερινή τους επαγγελματική χρήση. Υπάρχουν όμως πολλά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα και για το καθάρισμα των δεξαμενών νερού των ε, ε, πισίνων που χρησιμοποιούνται για κολύμβηση λοιπά. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα δύο κράτη-μέλη που έχουν συστήματα αδειοδότησης, τα αιτήματα για την αδειοδότηση ήταν πολύ περιορισμένα. Δεν κάνουμε λόγο για χιλιάδε, αλλά κάποιε μερικέ εκατοντάδε που ε, ζητούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια χημικά, τέτοιε χημικέ ουσίε. Δεν είναι τόσο αρνητικά λοιπόν τα πράγματα, όσο ίσω με μια πρώτη ματιά μπορεί να δημιουργηθεί εντύπωση. Και για του δύο καταλόγου. νομίζω υπάρχει σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των χημικών εκείνων όπου είναι εύκολο να υπάρξει όριο όσον αφορά τη συμπίκνωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι ασφαλή, αλλά όμω δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν έτσι, διότι έχουμε μεγάλο άλλους όγκους όπως ε, για παράδειγμα για το ασετόν ή για παράδειγμα το Εξαλέν που είναι πολίτες σε μικρούς κύβους ε, και υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την, ε, τα όρια. Λοιπόν, για οποιαδήποτε τέτοια χημική ουσία, αν υπάρχει ύποπτη συναλλαγή, όλα αυτά θα εφαρμόζονται. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ορισμός των ε, ύποπτων συναλλαγών πρέπει να προσδιοριστεί περισσότερο για να έχουμε μια σαφέστερη βάση. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι, ε, λαμβάνοντας υπόψη βάση παρατηρήσει παρατηρήσεις του επόπτη, Ευρωπαϊκού Επόπτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο λόγος ε, για τον οποίο δεν συμπεριλάβαμε αυτή την πτυχή στην πρόταση είναι ο λόγος της επικουρικότητας, το επιχείρημα της επικουρικότητας. Είναι θέματα που θα εφαρμοζόντουσαν σε όλα τα στοιχεία που ε, αποθηκεύονται ή συλλέγονται από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό ισχύει εκεί η αρχή της επικουρικότητας. Δεν είχαμε την δυνατότητα να βρούμε κάποια ε, περίπτωση όπου θα έπρεπε σε άλλο επίπεδο να γίνει αυτό. Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και η παρατήρηση του κυρίου Ντεγιόν για τις μικρές ε, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν είχαμε το σύστημα ε, καταχώρησης ε, σε ε, σχέση με το σύστημα αδειοδότησης και υπήρχε επιβάρυνση, όχι όμως προσπαθούμε να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές από κοινού ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν με εύκολο τρόπο να διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές. Αν κάποιος αγοράζει υδρογόνο, υπεροξίδιο του υδρογόνου και θα έπρεπε αυτό να είχε αναγνωριστεί ως επικίνδυνη συναλλαγή, ύποπτη συναλλαγή συναλλαγή δεν καταχωρήθηκε, δεν αναφέρθηκε με όλε τι γνωστέ επιπτώσει. Ευχαριστώ. Τώρα εσεί έχετε τον λόγο κύριε Μούλτερ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ όλου για τα σχόλια που έκαναν. Και θα λάβω υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Ματιέ σε σχέση με τις ε, απαντήσεις που δόθηκαν μπορούμε ίσως να δώσουμε και συνέχεια σε μεγαλύτερη ε, έκταση. Για όσα ανέφερε ο κ. Ντεγιόν ήδη στην πρώτη μου εισαγωγή είχα προαναφέρει ότι με τη βάση αυτά, αυτών που αναφέρονται για την προστασία προσωπικών δεδομένων ε, θα έχουμε και τροπολογίες για να καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσμα και όσον αφορά τον ορισμό των επικίνδυνων συμπεριφορών ή επικίνδυνων συναλλαγών όσον αφορά ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσπαθήσω να καταφέρω να βρω ένα καλύτερο ορισμό που θα είναι πιο αποδεκτός και για, το, για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Θα το προσπαθήσω λοιπόν. Ελπίζω λοιπόν τούτων λεχθέντων ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο γοργά, υλοποιώντα αυτή την σωστή καλή πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα έχοντας ακούσει και παρακολουθήσει τη συζήτηση, καλό και δίκαιο θα είναι να θέσουμε μια καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα είναι η Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011, 2011 το μεσημέρι, ναι, στις 12 το μεσημέρι. Θα είναι λοιπόν η αυτή η Παρασκευή, έτσι, η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Συμφωνούμε λοιπόν επ' αυτού. Εντάξει. Και συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας. Το σημείο 14 είναι αυτό. Η <clears throat> ενιαία διαδικασία για την ε, εργασία και την ε, άδεια αίτηση και άδεια παραμονής ε, εργασία στο υπαριθμό 14. Το έχουμε συζητήσει για αρκετό χρονικό διάστημα αυτό το θέμα και περάσαμε το σύνολο της διαδικασία ε, σε όλες τις φάσεις. Τώρα ας ακούσουμε το πώς έχουν τα πράγματα από την εισηγήτρια της Επιτροπής μας, τη συνάδελφο κυρία Βερονίκ Ματιέ θα τις δώσουμε τον λόγο λοιπόν. Δεδομένου ότι με τον τελευταίο τριμερή διάλογο που έγινε στις 22 Ιουνίου μια συμφωνία επετεύχθη. Μια συμφωνία επί της ουσίας Στη φάση μιας διαπραγμάτευσης για την πρώιμη, ας το πούμε έτσι, σε πρώτη ανάγνωση συμφωνία αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα και θέλουμε να ακούσουμε το τι συνέβη από τότε, πώς έχουν τα πράγματα από την εισηγήτρια, την κυρία Ματιό. Και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και από τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στον τριμερή διάλογο όσον αφορά το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μια και παρίστανται. Κυρία Ματιό, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, το είπατε κι εσείς ότι πολύ καιρό το συζητούμε αυτό το θέμα. Στον τελευταίο τριμερή διάλογο, στις 22 Ιουνίου, καταλήξαμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο και το σύνολο των πολιτικών ομάδων για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μετά από μακρόχρονες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, καταλήψαμε σε ένα ε, κείμενο που είναι αποδεκτό για όλους ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους πέντε στοιχεία παρέμεναν προς διαπραγμάτευση ε, καταφέραμε να επιτύχουμε μία περίοδο τεσσάρων μηνών ε, για τη χορήγηση της ενιαίας άδειας. Ε, καταφέραμε επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σήμερα για την άδεια εργασίας, είδος δραστηριότητας, τόπος άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ άλλων. Είναι μόνο μία επιλογή για τα κράτη-μέλη. Επιλέξαμε, επίσης την συμμετοχή του, σε επαγγελματική κατάρτιση, σε επιδόματα ανεργία. Διατηρήσαμε τη θέση μα επίση για το θέμα των συντάξεων, που πρέπει να είναι αντικείμενο ισότιμη μεταχείρισης και για του αλλοδαπού. Το Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες επιβεβαίωσε αυτήν την ε, ε, συμφωνία. Μόνο οι πίνακες αντιστοίχησης ε, παραμένουν εκκρεμείς, ειδικότερα ένα συγκεκριμένο σημείο, μια αιτιολογική σκέψη. Πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει μια οριζόντια λύση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Επίσης θα ήθελα να σας προτείνω ο πρόεδρός μας να μας στείλει, να στείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της Κορεπέρ λέγοντας ότι δεχόμαστε τη συμφωνία χωρίς τροπολογίες στο πλαίσιο μιας δεύτερης ανάγνωσης ε, με την επιφύλαξη εξέβρεση συμφωνία όσον αφορά του πίνακε αντιστοίχηση. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, και εγώ ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα την άποψη της πολωνική Προεδρίας. Όχι η κυρία Ανιές Κασκίβα, τότε ο κύριος που θα μας συστηθεί. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τόμας Τσιτρινόβιτς είναι το όνομά μου. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ματιέ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο καλοδέχεται, το, καλωσορίζει το αποτέλεσμα που επετεύχθη και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσει ο, αυτό το χαρτοφυλάκιο και όλη η διαδικασία των δυνατών πιο σύντομα. Ίσως αν αυτή η επιστολή που αναφέρατε φτάσει στο Συμβούλιο αυτήν την εβδομάδα, τότε θα συζητήσουμε στην Κορεπέ στις 20 Ιουλίου για αυτό το θέμα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είσαστε τόσο σύντομος και περιεκτικός. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιος θα ήθελε να παρέμβει, όχι. Εσείς, παρακαλώ εσείς κυρία. Λυπούμε, αλλά συνάδελφοι δεν είναι <laughs> ακόμα εδώ, είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα φτάσουν σε λίγα λεπτά. Δεν είναι παρόντα τα μέλη. Έχετε δίκιο ουσιαστικά, Νέγιο ο πρόεδρο. Ε, Στι 10.30 είχε καθοριστεί η συζήτηση, η εξέταση αυτού του θέματο. Κινδυνεύουμε τώρα να έχουμε κάποιο διάλειμμα που θα πρέπει να πάρει φρύση ακούσουμε από τον ε, διευθυντή της Eurojust που είναι ο ειδικό φιλοξενούμενος στο επόμενο σημείο που προβλέπεται για τις 11. Είμαστε πέντε λεπτά πιο μπροστά στο χρονικό πλαίσιο. Έρχεται έτσι, έρχεται λέτε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Νομίζετε ότι θα έρθει σε μερικά λεπτά ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής. Τι πιστεύετε. Το ελπίζω. Διότι βρίσκεται μάλλον καθοδόν. Είναι κάπως δύσκολο να έχουμε την ε, άμεση επαφή. Δεν βλέπω, λέει ο Πρόεδρος, κάποια άλλη μέλη που να θέλουν να παρέμβουν για αυτό το συγκεκριμένο θέμα ή σε αυτή τη φάση της συζήτηση. Ε, τότε λοιπόν ας σας αναγγείλω σε αυτή την περίπτωση ότι σε σχέση με αυτό το θέμα, όπως προαναφέρθηκε, εγώ θα αποστείλω ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, μια επιστολή στον πρόεδρο της Κορεπέρ όσον αφορά το σημείο 18 κοινή δήλωση για πρακτικές ε, ε, συμφωνίες για τη διαδικασία συναπόφασης για ενημέρωση όσον αφορά την συμφωνία ε, όσον αφορά τον τριμερή διάλογο. Εν πάση περιπτώσει σωστό και δίκαιο είναι να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να διακόψουμε σύντομα για μικρό διάστημα αυτή τη συνεδρίαση πρωτού συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο καθώς ο διευθυντής της Eurojust θα πρέπει να προσέρθει σε κάποια λεπτά. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε στη συνέχεια να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο, δηλαδή να ακούσουμε σε σχέση με την ετήσια έκθεση της Eurojust για το 2010. 15 λεπτά καλά είναι μέχρι να έρθει 15 λεπτά, είναι τεταρτάκι μέχρι να προσέλθει ο Γενικός Διευθυντής. Συμφωνείτε? Εντάξει λοιπόν. Ε, λοιπόν, θα διακόψουμε για ένα τεταρτάκι. Διακοπή. Ευχαριστώ.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 Dear colleagues. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, We are still for once ahead of time. Μία ακόμη φορά Είμαστε νωρίτερα σε σχέση με το πρόγραμμά μας, 15 ολόκληρα, 15 ολόκληρα λεπτά. Όμως είναι εδώ ο πρόεδρος της Eurojust, ο κύριος Άλεντ Williams, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω θερμότατα θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της Eurojust για το 2010. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που απολαμβάνουμε την παρουσία του κυρίου Williams εδώ στην Επιτροπή μας. κάτι το οποίο δείχνει την ε, συνεργασία που θα έχουμε ως Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτό το αξιότιμο όργανο, τη Eurojust, που αφορά τη δικαιοσύνη και τα, τις εσωτερικές υποθέσεις, είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ε, μελλοντικής ανάπτυξης ε, του ε, χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, από το 2002, κάθε προσπάθεια που έχει γίνει από τη Eurojust προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ των ε, διαφόρων φορέων που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου έχει επιβεβαιώσει ακριβώς την ανάγκη ύπαρξη τέτοιας, ύπαρξης μια τέτοια συνεργασίας. Οπότε θα ακούσουμε την παρουσίαση της τελευταίας έκθεσης της Eurojust του 2010 και μετά θα γίνει συζήτηση. Um, κύριε Βίλιαμς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για, αυτά τα καλά σας λόγια και θα ήθελα ευθύ αμέσω να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και ε, προνόμιο για τη Eurojust ε, να μπορεί να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση ε, για το 2010 στην Επιτροπή σας. Είναι ιδιαίτερος σημαντικό για την Eurojust γιατί Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, ο οποίος ε, ενισχύθηκε ε, στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας ε, σε σχέση με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας. Οπότε εμείς βλέπουμε την ετήσια έκθεσή μας ως κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να χρησιμεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο καθήκον αυτό της αξιολόγησης των, ε, των δραστηριοτήτων μας. Οπότε, όπως είπε και ο πρόεδρος ε, κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης των δεσμών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα εθνικά κοινοβούλια, η Eurojust ε, πάντοτε ε, ήταν έτοιμη και ε, ευγνώμων να προσέλθει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σας. Κατά τη διάρκεια του 2010, εκπρόσωποι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ επίσης ήρθαν στη Χάγη στις ε, εγκαταστάσεις της Eurojust ε, και είχαμε συζητήσει σε σχέση με το τρίο της Προεδρίας, όπως επίσης ε, και με τις οδηγίες που αφορούσαν ειδικότερα την, τα θέματα εισαγγελία και άλλου είδου ζητήματα στην Ευρωπαϊκή, στο χώρο δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δεν μπορεί να είναι ένα πλήρες ε, εργαλείο αξιολόγησης η έκθεση αυτή. Νομίζω όμως ότι μπορεί πραγματικά να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την αξιολόγηση στην οποία πρέπει να προβεί. Αυτό που θα ήθελα να κάνω, αν μου το επιτρέπει ο ε, Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίασής μου, είναι να ασχοληθώ με τρεις κύριες θεματικές ενότητες που πιστεύω ότι προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του 2010. Η πρώτη θεματική ενότητα έχει να κάνει με την απειλή του ε, διασυνοριακού εγκλήματος. Η δεύτερη ε, θεματική ενότητα, κάπως πιο τεχνική, είναι η μετάβαση από την αμοιβαία νομική ενίσχυση ε, προς την αμοιβαία αναγνώριση κάποιων αποφάσεων στην, ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον, ε, κάτι που επίσης προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Eurojust για το 2010 είναι κάποιες, κάποια ενδεχόμενα κάποιες ενδεχόμενες κάποια πορεία που μπορούμε να έχουμε Κάπω πιο ενισχυμένη προς το χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Οπότε α μιλήσω πρώτα για το πρώτο θέμα που ανέφερα, την απειλή από το διασυνοριακό ε, έγκλημα και τα στοιχεία που έχουμε στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης το 2010. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να σας φαίνεται αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί μια ακόμη φορά και αυτό είναι η απειλή ε, στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το διασυνοριακό έγκλημα δεν έχει μειωθεί δεν έχουμε καταφέρει να ε, εξαλείψουμε ε, τον αντίκτυπό της ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της, του 2010 με πάνω από 1.400 υποθέσεις οι οποίες μας παραπέμπονται είτε από τους, είτε από τους εταίρους μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Όλαφ και η Ευρωπόλ είτε ε, και από ε, τα κράτη-μέλη. Ενδεχομένως ε, να εξηγείται αυτή η αύξηση των υποθέσεων διασυνοριακού εγκλήματος, να μην είναι η αύξηση αυτού, αλλά το γεγονός ότι μετά από 10 χρόνια ύπαρξής της η Eurojust είναι πλέον πιο γνωστή στις αρμόδιες αρχές και σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και σε επίπεδο εθνικό. Ωστόσο, ε, πιστεύω ότι δεδομένης της σταθερής αύξησης για ε, ενίσχυση από την Eurojust, να σας ε, πω για παράδειγμα ότι το 2002 είχαμε να ασχοληθούμε με, δύο, με 200 υποθέσεις, με συγχωρείτε. Πέρσι είχαμε 1.400 υποθέσεις των οποίων έπρεπε να επιληφθούμε. Βλέπετε ότι είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Δεν έχει μειωθεί λοιπόν η απειλή από το διασυνοριακό έγκλημα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ο αριθμός των συντονιστικών συνεδριάσεων ε, που ε, γίνεται ε, με τη Eurojust έχει αυξηθεί επίσης. Πάνω από 140 τέτοιου είδους συνεδριάσεις υπάρχουν και νομίζω ότι αυτό δείχνει την προστιθέμενη αξία είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι ε, αρκετά εμφανές πλέον και ορατό στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Η ιδέα της ε, συνεδρίασης της συντονιστικής είναι πάρα πολύ απλή. Νομίζω ότι πρέπει να πω όμως ότι είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματική μια τέτοιου είδους συνεδρίαση γιατί συγκεντρώνει, δεν είναι βέβαια πάντα εύκολο, σε επίπεδο Eurojust ε, ε, ανακριτές, ε, εισαγγελείς, δικαστές που ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις στα κράτη-μέλη, συναντιούνται με εμπειρογνώμονες της Eurojust, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι μπορούν να μιλήσουν ο καθένας στη γλώσσα του με υψηλό επίπεδο διερμηνίας και άλλων και άλλης τεχνικής αρρωγής που τους ε, παρέχετε, Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές και, και τακτικές όσον αφορά την ε, ε αντιμετώπιση τέτοιου είδους διαστηνοριακών υποθέσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, πολύ σύντομα, ε, το οποίο αναφέρεται και στην ετήσια έκθεσή μας. πρόκειται... Την υπόθεση Lost Boy που μας έδωσε τη δυνατότητα να ε, δούμε όλα τα στοιχεία ε, συνεργασία συντονισμού στο πλαίσιο της Eurojust θα πρέπει να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε ε, μας έδειξε αυτή η υπόθεση ε, τους ε, εισαγγελείς ε, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. επίξε και μία υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και στο διαδίκτυο. Αφορούσε μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία. Κάποιος συνελήφθη στην Νορβηγία, κατηγορούμενος για κακοποίηση ενός παιδιού στην Νορβηγία ε, εκτός από τους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών, ε, η Eurojust ε, έχει και κάποιους εκπροσώπους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Κροατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την, υπόθεση υπήρξε μία σύλληψη ενός υπόπτου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ε, υπήρξαν κάποια στοιχεία στο σπίτι του και όταν ε, έψαξαν στο σπίτι του είδαν εκτός ε, από κάποιες ε, φωτογραφίες που επιβεβαίωναν ε, κάτι τέτοιο, κάποιες επαφές και κάποιες, κάποια καταγραφή συνομιλιών που είχε στο διαδίκτυο συγκεκριμένος ύποπτος με διάφορους άλλους συνεταίρους του σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επτά κράτη-μέλη συνολικά αφορούσε η υπόθεση αυτή και μάλιστα το δίκτυο αυτό έφτανε μέχρι τις Ηνωμένε Πολιτείες, το Αφγανιστάν και τη Βραζιλία. Το γεγονός λοιπόν αυτής της ανταλλαγής ε, μεταξύ των ε, ε, εγκληματιών αυτών και μέσω του διαδικτύου αναφέρθηκε ε, στη δικαστική αρχή της Νορβηγίας ε, ε, και στην, στους εκπροσώπους μας εκεί της Eurojust και ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Eurojust και μιλώ για τις χώρες που των οποίων υπήκοοι συμμετείχαν στην υπόθεση αυτή της ε, μετάλλευσης των παιδιών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε όλα τα στοιχεία που υπήρχαν ε, και προσπαθήσαμε να δούμε ε, το, προσπαθούσαν οι άνθρωποι αυτοί να ε, δουν σε ποιες χώρες ήταν ευκολότερη αυτή η εκμετάλλευση των παιδιών ε, και προσπαθήσαμε τότε να οργανώσουμε μια συντονιστική συνεδρίαση σαν αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως όλων των κρατών μελών τις οποίες έπληξε ε, η υπόθεση αυτή και βέβαια των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες προέρχονταν οι υπόλοιποι ύποπτοι και διαπιστώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ απαραίτητο να καταλήξουμε σε αποφάσεις. Ε, έχουμε τη δυνατότητα ως Eurojust να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ποια χώρα έπρεπε να επιληφθεί τη υποθέσεως αυτής. Γιατί, όπως είπα, είμαστε εμπειρογνώμονε ε, στην επίλυση ε, συγκρούσεων ε, δικαιοδοσιών. Όταν ένα κράτος μέλος λέει ότι εκείνο είναι αρμόδιο να αναλάβει την υπόθεση, κάποιο άλλο κράτος μέλος λέει ότι και αυτό είναι αρμόδιο να αναλάβει την υπόθεση αυτή. Υπήρξε μια, υπήρξαν διάφορες επιπλοκές, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την υπόθεση μία εκ των οποίων ήταν ότι κάποιος από τους υπόπτους ε, είχε έρθει από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε αναλάβει μία θέση σε κάποιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν υπήρχε κανένα προηγούμενο μητρό ποινικό για τον άνθρωπο αυτό, ε, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κρατος μέλος. Και για να ε, και, το, το χειρότερο ήταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ε, που ήταν ε, κατηγορούμενος ε, για παιδική εκμετάλλευση συμμετείχε και σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που, λέγεται «Σώστε τα παιδιά». Οπότε ήταν, συμμετείχε λοιπόν σε αυτή τη φιλανθρωπική οργάνωση, ήταν μέλος αυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα και ήταν ένας άνθρωπος που επιδιδόταν σε αυτήν την πρακτική της παιδικής εκμετάλλευσης. Οπότε Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ε, ε, παρακολουθηθεί αυτός ο άνθρωπος ε, γιατί δεν, υπήρξε, δεν υπήρχε προηγούμενο ποινικό μητρό και δεν υπήρχε καμία υποψία εναντίον αυτού του ανθρώπου. Όμως η Eurojust κατάφερε να ξεκινήσει ε, μια ε, ανακριτική έρευνα για το θέμα αυτό κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ε, και σας το λέω για να σας δείξω πόσο σημαντική ήταν η συμβολή της Eurojust εν προκειμένου. Μετά λοιπόν από την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων που είχαν να κάνουν με το πώς έπρεπε να πλαισιωθούν τα ευρωπαϊκά συντάλματα, εντάλματα συλλήψεως, σε ποια κράτη-μέλη έπρεπε να υπάρξουν τέτοιου εντάλματα, τι διαδικασία διαδικασία έπρεπε να ακολουθηθεί ε, όταν μια διαδικασία είχε ξεκινήσει ήδη σε ένα άλλο κράτος μέλος, αλλά έπρεπε παράλληλα να γίνει και στο κράτος μέλος στο οποίο υπήρχαν οι υπόλοιποι ύποπτοι. Ε, όλες, ε, όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα 70 παιδιά να διασωθούν από την παιδική εκμετάλλευση μέσω της συντονισμένης αυτής διαδικασίας της Eurojust και συνελήφθησαν πολύ υποπτοί στο πλαίσιο αυτού του, ε, αυτής της προσπάθειας από το δίκτυο αυτό και ο άνθρωπος αυτός που δούλευε για τη φιλανθρωπική οργάνωση στο Λονδίνο που λεγόταν Save the Children, σώστε τα παιδιά. Οπότε ο άνθρωπος ε, αυτός ε, είχε μια διοικητική θέση στη φιλανθρωπική οργάνωση, δεν ερχόταν σε επαφή άμεση με τα παιδιά, δεν υπήρχε δηλαδή άμεση ε, ε, επαφή του ανθρώπου αυτού με τα παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός ε, φυλακίστηκε για πολλά χρόνια λόγω των δραστηριοτήτων που ορισμένες από αυτές ήταν πραγματικά φρικτές εκμετάλλευσης παιδιών ενός έτους. Και αυτό σας το λέω για να σας δείξω απλώς ε, την, ε, το είδος της εργασίας ε, την οποία κάνει η Eurojust και επιτρέψτε μου να σας πω πάρα πολύ σύντομα να επανέλθω και να αναφερθώ στην απειλή του οργανωμένου διασυνοριακά εγκλήματος που η Eurojust αντιμετωπίζει. Οι περιπτώσεις που έχουμε στην ετήσια έκθεση καταδεικνύουν ότι όσον αφορά δύσκολες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και δύσκολες περιπτώσεις που διαβιβάζονται σε εμά κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν απλές λύσεις απλά. Έχουμε κάτι, δηλαδή η αναλογία είναι απάτες ακόμα και το πλήσιμο χρήματος είναι οι περιπτώσεις εκείνε όπου έχουμε τον μεγαλύτερο συντονισμό, τι περισσότερε συντονιστικέ διασκέψεις. Ακολουθούνται από τις περιπτώσεις ε, για ναρκωτικά. Από αυτές, από τις 140 συντονιστικέ διασκέψεις, 54 ενέπλεκαν είτε την διαφθορά είτε το πλήσιμο χρήματος και είχαμε και περίπου 40 που αφορούσαν το εμπόριο ναρκωτικών. Ένα ξεχωριστό στατιστικό στοιχείο των ε, εκθέσεων είναι ότι στις συντονιστικές αυτές διασκέψεις, συνεδριάσεις που έχουμε στη Eurojust πάνω από 90% εμπλέκουν τα εγκλήματα που θεωρούνται ως ιδιαίτερες απειλές κατά των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρωταρχικής προτεραιότητας σε εγκληματικές περιπτώσεις που πρέπει να καταπολεμηθούν. Και όπως χαρακτηρίζονται έτσι ακριβώς οι περισσότερες συντονιστικές μας συνεδριάσεις αφορούν αυτές τις προτεραιότητες εμπόριων ανθρώπων, διαφορετικού είδους απάτες, κυβερνοέγκλημα και άλλου είδους εγκλήματα κατά της ε, κοινωνίας που διαπράττονται τα εγκλήματα αυτά από το οργανωμένο έγκλημα και τους εκπροσώπους του. Σωστό είναι να πει κανείς ότι η απειλή λοιπόν <clears throat> στους πολίτες της Ευρώπης από διασυνοριακό έγκλημα <clears throat> δεν μειώνεται. Η απειλή δεν μειώνεται. Και αυτό καταδεικνύεται από τον αριθμό των περιπτώσεων που διαρκώς αυξάνεται στη Eurojust. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, ας στραφώ σε μια άλλη πτυχή της ετήσιας έκθεσης. Και αυτή αφορά αυτό που πιστεύω εγώ ότι ίσως αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από εμά μια επαναστατική αλλαγή στην προσέγγιση σε σχέση με την δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η αλλαγή από την αμοιβαία δικαστική νομική σύνδρομη στην αμοιβαία αναγνώριση. Επαναστατική αλλαγή αυτή για την αμοιβαία αναγνώριση. Διότι αντικαθίσταται η νομική συνδρομή από την νομική αναγνώριση. Και αυτό πάει 10 χρόνια, πάει πίσω στο Τάμπερε, συμφωνία του Τάμπερε και πρόσφατα εφαρμόζεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και αντανακλάται στο άρθρο 82 που αναφέρει την αμοιβαία αναγνώριση ως τη βασική αρχή επί της οποίας θα πρέπει να λειτουργεί η δικαστική συνεργασία. Όμως πιστεύω στην θεωρία τουλάχιστον είναι κάτι που έχει τεράστια σημασία για τη διάθεση τη δόμηση ενός τομέα μιας περιοχής ε, ελευθερίας, δικαιοσύνης ε, και ε, δικαίου και έχουμε και δημοκρατίας. Έχουμε το σύστημα αιτήσεων και ετοιμάτων μια κρατική αρχή ζητά από μια άλλη ανεξάρτητη κυρίαρχη νομική αρχή για συνδρομή. Μετακινούμαστε από αυτό, μετατιθέμεθα από την αναγνώριση των νομικών πραγμάτων και αποφάσεων αμοιβαία από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, εξίσου σημαντικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της δράσης για τον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, την περιοχή αυτή είναι μετακινούμαστε από ένα κεντρικά σχεδιασμένο και κεντρικά, ε, ε, κεντρικό σύστημα σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Και έτσι δεν θα έχουμε στο μέλλον στενοπούς και προβλήματα όπως αυτά που είχαμε στο παρελθόν για τη δικαστική συνεργασία. Το να παίρνει κανείς εντάλματα ή εντολές για έρευνα, σε κατοίκον έρευνα, σε έλεγχο λογαριασμό τραπεζικών ή και ε, εντάλματα σύλληψης από τη διαβίβαση από κεντρικές αρχές στο μέλλον θα έχουμε αποκεντρωμένο σύστημα λειτουργίας. Μία δικαστική αρχή σε ένα κράτος μέλος θα είναι σε θέση, θα μπορεί να ανταποκρίνεται και να διαβιβάζει άμεσα το αίτημά της στις δικαστικές αρχές άλλου κράτους μέλους και άμεσα θα εκτελείται η εντολή αυτή η πτυχή, αυτή η μετάθεση, η μετακίνηση στην αμοιβαία αναγνώριση λέει η ετήσια έκθεση και τονίζει στο έργο της Eurojust ίσως ακριβώς το πιο επιτυχές στοιχείο και εργαλείο της αμοιβαίας αναγνώρισης που είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. European Arrest Warrant. Από τις χιλιάδες και τόσα ε, εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 αυτή τη στιγμή δεν έχω τα στοιχεία το 2010 λυπάμαι γι' αυτό, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αύξηση από τις 14.000 εντάλματα του 2009. Όσον αφορά λοιπόν τη Eurojust, εμείς θεωρούμε και ισχυριζόμαστε ότι αυτό μπορεί να περιγραφεί ως ένα χρήσιμο και πραγματικά ένα σημαντικό εργαλείο, διασφαλίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης θα λειτουργούν στην πρακτική εφαρμογή και θα είναι αποτελεσματικά. Έχουμε αιτήματα να ε, εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν δυσκολίες σε περίπου 280 περιπτώσεις. Δηλαδή κάπου 20% των περιπτώσεων που διαβιβάζονται σε εμάς στην Eurojust αφορούν δυσκολίες που αφορούν επίλυση προβλάτων όσον αφορά θέματα ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψη. Ένα απλό παράδειγμα να σας δώσω. Κάτι που απαιτείται να πράττουμε εμεί να κάνουμε υπό το πρίσμα τη απόφαση πλαισίου για το ευρωπαϊκό ενταλμα σύλληψης. Τι συμβαίνει αν ένα άτομο συλλαμβάνεται σε ένα κράτο μέλο και διαπιστώνεται ότι περισσότερα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να τον συλλάβουν και να τον προσαγάγουν σε δικαιοσύνη, σε δίκη. Έχουμε πολλαπλά λοιπόν δικαστικά δικαστικά εντάλματα και άμεσα τριβές δικαστικές. Ποιος θα πάρει αυτόν τον ε, καταζητούμενο. Και στην ετήσια έκθεση εφέτος, όταν ένα άτομο συλλαμβάνεται για παράδειγμα από τις βελγικές αρχές και διαφαίνεται και διαπιστώνεται ότι αυτό το άτομο καταζητείται όχι μόνο στο Βέλγιο για παραπτώματα και αδικήματα, αλλά και στη Γερμανία και στην Αυστρία και όπου τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για αυτόν. Ε, αυτό το άτομο ε, συνελήφθη, κρατήθηκε και είναι θέμα ταχύτητας άμεσης επίλυσης αυτών των δικαστικών τριβών, αυτών των προβλημάτων σε σχέση με τις γερμανικές και αυστριακές αρχές των ενταλμάτων σύλληψης, μια και αυτός ε, είχε συλληφθεί από το Βέλγιο και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορείτε να φανταστείτε ποιες δυσκολίες αναφύονται δεν έχουμε ένα σώμα σαν την Eurojust να επιλύει αυτά τα προβλήματα όπου σε αυτή την περίπτωση ακριβώς το θέμα επιλύθηκε μέσα σε 72 ώρες νομίζω όλες και όλες και επιλύθηκε με πολύ απλό και άμεσο τρόπο κιόλας. Οι βελγικές αρχές ήρθαν σε επαφή με το εθνικό μέλος της Eurojust, εκείνη η κυρία ήρθε σε επαφή με τον γερμανό και αυστριακό εταίρο συνδέσμους στη Eurojust, συζήτησαν την περίπτωση πάντα φυσικά με επαφή και σε επαφή με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών, τις αρμόδιες κρατικές εθνικές αρχές. Και ήταν πολύ εύκολο και άμεσο να επιτευχθεί μια λογική επίλυση των προβλημάτων αυτών των αντιφατικών στοιχείων των ευρωπαϊκών ενταλμάτων είχαν εκδοθεί για σχετικές και συναφείς κατηγορίες και αδικήματα. Φανταστείτε μια κατάσταση αν δεν υπήρχε η Eurojust και τις δυσκολίες που θα πέραν να μπορέσει να ταυτοποιηθεί μια, ε, ένα άτομο σε σχέση με το τι θα έπρεπε να συμβεί με αυτόν. Δεν θα ήταν εύκολο να υπάρξει συνεννόηση και σε μια κοινή γλώσσα ακόμα και τέτοια απλά πράγματα. Αυτή η παρέμβαση σήμαινε ότι οι δυσκολίες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταμα Σύλληψης πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν και άλλες πολλές δυσκολίες που δεν θα επισέλθω σε αυτές τώρα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Υπάρχουν πολλές και άλλες δυσκολίες εμπλέκουν πράγματα όπως δίκες ερήμην των κατηγορουμένων, τη απουσία τους. Τι κάνει δηλαδή κανείς όταν κάποιος καταδικάζεται ερήμην σε κάποιο κράτος μέλος. Δεν είναι παρόν στη δίκη, μετά όμως ε, φεύγει, δραπετεύει σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και εκείνο το κράτος έχει δυσκολία να παραδώσει, να εκδώσει αυτό το άτομο χωρίς εγγυήσεις από το αρχικό κράτος μέλος για ε, εγγυήσεις για δίκαιη δίκη και τα λοιπά. Τέτοιου είδους προβλήματα και περιπλοκές. Υπάρχει επιπρόσθετα όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ένα συγκεκριμένο νέο στοιχείο, μέσο ή εργαλείο που βρίσκεται υπό συζήτηση και όπου εκεί έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η Eurojust και που αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή μας και είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερευνών για μας ε, στην διασυνοριακή δικαστική συνεργασία αυτό το μέσο, το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας ή ερευνών μπορεί να δημιουργήσει, να συναποτελέσει μια επανάσταση στον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή ε, το ένταλμα αυτό εξατάζεται ακόμα από τα κράτη-μέλη μέσα στο πλαίσιο του πλαισίου του Συμβουλίου. Είναι όμως μια πρόταση που σύντομα, προσεχώς, θα έρθει, θα προσέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εξέταση και έγκριση. Στην ουσία του θα είναι, ας το πω έτσι, θα συγχωνεύει και θα συγκλίνει όλα τα μέσα για την δικαστική συνεργασία σε αυτό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συναποτελεί μία πάγια βάση, ένα κωδικοποιημένο πάγιο μέσο που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε δυσκολίες που υπάρχουν στην πρακτική εφαρμογή συχνά. Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές πιθανές δυνατότητες και τρόποι κάποιος να προχωρήσει ζητώντας δικαστική συνεργασία από ένα άλλο κράτος μέλος. Τι θα κάνει αυτός πάει και θα έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, θα χρησιμοποιήσει τη σύμβαση του 1959, τι άλλο θα κάνει, θα χρησιμοποιήσει τη σύμβαση του 2000 τόσο ε, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σχετικό πρωτόκολλο για αυτό το μέσο έχει δικαίωμα αυτό να κάνει και να χρησιμοποιήσει αυτό. Θα χρησιμοποιήσει τη σύμβαση Σέγγεν, τέτοιου είδους προβλήματα. Όλα αυτά δημιουργούν πρακτικά προβλήματα και τριβές για τις διοκτικές αρχές, τους εισαγγελείς, τους δικαστές, τις αρχές ε, εφαρμογής του νόμου, τις δικαστικές αρχές όταν έρχεται η ώρα να καταπολεμηθεί άμεσα το οργανωμένο έγκλημα και οι πρόσωποι του. Αυτή η συγκεκριμένη πρόταση που σύντομα προσεχώς θα έρθει στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εξέταση και έγκριση είναι κάτι που έχει τεράστια σημασία και κάτι που η Eurojust συνεισέφερε η ίδια στη συζήτηση για ορίμανση αυτών των προτάσεων και ελπίζουμε ότι θα είναι μια πρόσκληση έτσι σε σχέση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ υπό τους ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις να συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση, στη συζήτηση που θα διεξαχθεί για αυτό το μέτρο από πλευρά τη. Στη συνέχεια, αν μου επιτρέπετε σύντομα, να έρθω στο τελευταίο ζήτημα, στο τελευταίο θέμα που θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με την ετήσια έκθεσή μα. Και αυτό είναι οι τρόποι με του οποίου η διασυνοριακή δικαστική συνεργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί στο μέλλον θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ομολογήσω και εξ ονόματος της Eurojust αυτό ότι έχουμε στο παρελθόν ίσως επικεντρωθεί περισσότερο στις εργασίες μας στις πρακτικές μορφές των περιπτώσεων σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και δεν συναγάγαμε τόσο πολύ συμπεράσματα και μαθήματα από αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα όμως το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό ότι πρέπει να γίνει και δεν έγινε και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να περιγράψουμε να γίνουμε ένα κέντρο πραγματογνωμοσύνης και γνώσης όσον αφορά την δικαστική συνεργασία με συγκεκριμένα μαθήματα και ε, συμπεράσματα που σας συναγάγουμε. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιπτώσεων, συγκεκριμένες περιπτώσεις από τις οποίες είτε έχει ταυτοποιήσει ή έχει εντοπίσει ή έχει προτείνει λύσεις η Eurojust. Μία περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό είναι εκείνη όπου η Eurojust ε, εντόπισε το πρόβλημα αλλά θα έπρεπε να εξετάσει τα θέματα των νομοθετών των νομοθετικών αρχών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για μια επίλυση του προβλήματος. Αυτό αφορά την ε, συλλογή πληροφοριών από τα κράτη-μέλη πληροφοριών. Είναι κάτι το κοινότοπο, κοινό από ό,τι γνωρίζετε, τα τηλέφωνα των εγκληματιών ε, να παρακολουθούνται. Υπάρχουν όμως κανόνες και κανονισμοί που θεσπίζονται και που στη σύμβαση του 2000 έχουν εγκριθεί για την ε, αμοιβαία νομική δικαστική αρρωγή μεταξύ κρατών μελών. Τι θα γίνει αν ένας έμπορος ναρκωτικών πάει τώρα από το Βέλγιο, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Εντάξει, και τώρα χρησιμοποιεί εκεί το κινητό του τηλέφωνο ακολουθώντας εγκληματικούς σκοπούς και στόχους για να μπορέσει να αγοράσει ή να πουλήσει ναρκωτικά ενώ βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι κανονισμοί και οι κανόνες τι λένε αυτή τη στιγμή. Το κράτος μέλος που ενδιαφέρεται το Βέλγιο σε αυτή την περίπτωση που ενδιαφέρεται στη δίωξη αυτού του ατόμου που λειτουργεί τώρα και δρά στη Γαλλία. Οι κανόνες λένε ότι είναι αναγκαίο αυτό το κράτος μέλος να ειδοποιεί έγκαιρα το ε, κράτος μέλος υποδοχής, τη Γαλλία δηλαδή, ώστε εκείνο να παρέμβει και να παρακολουθήσει την τηλεφωνική συνδιάλεξη στην επικράτειά του, μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Ωραία όλα αυτά, όταν έχει συνειδητοποιήσει και γνωρίζει ένα κράτος μέλος τον στόχο της δράσης στην επικράτειά του. Τι γίνεται όμως αν έχουμε τις σημερινές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Πολύ συχνά τι συμβαίνει. Το κράτος μέλος που, είναι, που στοχοθετεί αυτόν τον εγκληματία δεν θα παρακολουθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν θα γνωρίζει ότι βρίσκεται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους ο εγκληματίας. Στην πρακτική εφαρμογή, στην δίωξη, στις διοκτικές δράσεις και στο δικαστικό επίπεδο είναι ε, αυτόματα καταγράφονται, μαγνητοφωνούνται λέει αυτές οι συνδιαλέξεις και αυτόματα αυτό το υλικό θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην δίωξη σε μια ε, ανακριτική δράση ή όχι. Αυτό αμέσως όμως θέτει πιθανά προβλήματα όσον αφορά την, το αποδεκτό στα δικαστήρια ως αποδεικτικών στοιχείων, ως τεκμηρίων αυτών των στοιχείων. Οι Βέλγοι αξιωματούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες μαγνητοφωνημένες συνδιαλλαγές συνδιαλέξει στην επικράτεια ενό άλλου κράτου μέλου. Θα μπορεί να αντιμετωπίζουν θέμα μη αποδεκτού, μη παραδεκτού υλικού. Και έτσι σε αυτή την περίπτωση εδώ η νομοθεσία δεν παρέχει λύση αυτόματα για αυτέ τι αυτόματε καταγραφέ ε, μαγνητοφωνήσει συνδιαλέξεων και για την χρήση αυτού του υλικού άμεσα. Μπορείτε αμέσω να δείτε ότι αυτό δημιουργεί ένα φάσμα για διάφορα επιχειρήματα που μπορούν εδώ να εγερθούν αν μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί και μάλιστα εσκεμμένα ή εν γνώση παραβιάζοντας τη σύμβαση. Τέτοιου είδου θέματα είναι εξειδικευμένα αυτά που η Eurojust έχει ταυτοποιήσει και ταυτοποιεί. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν κάτι το οποίο θα απαιτούσε στη συνέχεια νομική επίλυση του προβλήματος στο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου και εξέταση. Όμως σε γενικού όρους όσον αφορά το μέλλον μπορούμε να πούμε ότι η ετήσια έκθεση νομίζω αναφέρει αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτα, την σημασία, σπουδαιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αξιωματούχους και υπαλλήλους της Eurojust και το τονίζουμε αυτό επανειλημμένα στην ετήσια εκθεσή μας. Ιδιαίτερα έχει μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία για μας υπό το άρθρο 13, διότι υπό το άρθρο 13 της νέας απόφασης της Eurojust που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 4η Ιουνίου 2011, εφέτος, πολύ πρόσφατα δηλαδή, υπάρχει άμεση υποχρέωση από τα κράτη-μέλη να παράσχουν στη Eurojust ουσιαστικά λεπτομέρειες οποια, οποιασδήποτε περίπτωσης διασυνοριακής που εμπλέκονται και γνωρίζουν για αυτήν και όπου ουσιαστικά τρία κράτη-μέλη θα εμπλεκόντουσαν σε τριγωνική σχέση. Υπάρχει υποχρέωση αμέσως να αποστέλλονται πληροφορίες στη Eurojust σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό έχει ζωτική σημασία για μας. Αν δεν πάρουμε τέτοιου είδους πληροφορίες δεν είμαστε σε θέση να έχουμε θετικά αποτελέσματα, πρόσθετη αξία από τις έρευνες. Επιπρόσθετα όσον αφορά αυτό το στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών και ανταλλαγής δεδομένων, η Eurojust όπως αναφέρεται στην έκθεση κάνει σημαντικές συνεισφορές όσον αφορά τις δράσεις της Europol. Ιδιαίτερα παρέχουμε ένα δικαστικό πλαίσιο και προοπτική στην αξιολόγηση απειλών και δίωξη των εγκληματιών καθώς επίσης και τις περιπτώσεις όσον αφορά δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και τρομοκρατικές ή εγκληματικές. Αυτού του είδους ε, οι δράσεις έχουν κέρια σημασία ως στοιχεία για να βελτιωθεί η προστασία των πολιτών από το διασυνοριακό έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη μείζον πτυχή η οποία απορρέει από αυτή την έκθεση θα έλεγα ως φάσμα που έχει δυνατότητα δυνατότητες ε, βελτιώσεων στο μέλλον είναι η εταιρική σχέση ήδη προηγούμενα υπενήχθηκα εν παρόδο στην ανάγκη να υπάρχει αυτή η εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρήχαμε, ε, ε, είχαμε παράσχει υλικό για μελέτες όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο πρόσφατα ε, όσον αφορά την ίδια την έκθεση για την μελέτη για το πώς το οργανωμένο έγκλημα δρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει κατάχρηση των κονδυλίων ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται απάτες με τη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί η εταιρική σχέση σε λειτουργικό επίπεδο με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σχέση μας με Europol, την Europol. Αυτή τη στιγμή από τις 140 τόσες συναντήσεις συντονισμού η Europol, η Ευρωπόλ σε ένα τρίτο είναι παρούσα και συμμετέχει. Αξιόλογο αυτό το ποσοστό ως αριθμητικό μέγεθος. Μπορεί όμως να βελτιωθεί αυτό. Και έχουμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Χάγη να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν στενότερα μεταξύ μας. Μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις με την Ευρωπόλ έχουν βελτιωθεί. Όμως ακόμα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, ακόμα πιο πολύ. Και όταν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα για προτάσεις για κανονισμούς προτάσεις κανονισμού και για την Eurojust και για την Europol, Europol που κατανοώ ότι μπορεί να υπάρξει το θέμα της εξέτασης αυτών των θεμάτων είτε φέτος είτε του χρόνου. Σίγουρα όσον αφορά εμάς τους ίδιους ως Eurojust ελπίζουμε ότι θα είναι προτάσεις κανονισμού που θα εξεταστούν ε, για του χρόνου. Διότι πιστεύω εγώ και απορρέει και από την ίδια την έκθεση ότι είναι σημαντικό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο αυτές οι προτάσεις να εξετάζονται από κοινού σε νομοθετικό πλαίσιο προτάσεις για κανονισμούς. Ιδιαίτερα λόγω της φύσης ε, του συσχετισμού μεταξύ Eurojust και Europol, Europol που πρέπει να ενισχυθεί η σχέση αυτή νομοθετικά με κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λειτουργικά συνεργαζόμαστε και λειτουργούμε πολύ καλά ο ένας με τον άλλον. Όμως σε σχέση με την απόφαση για την Ευρωπόλ εμείς αντιμετωπιζόμαστε ως τρίτος ε, εμπλεκόμενος, τρίτος εταίρος. Δεν έχουμε αν θέλετε μια προνομιακή σχέση ε, ιδιαίτερης, ε, ε, ιδιαίτερα ευνοϊκής αντιμετώπισης ή προτίμησης σε σχέση με την Europol, την Ευρωπόλ έναν προτιμησιακό εταίρο, όχι την Ευρωπόλ, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, European Judicial Network. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη στο μέλλον αυτό το στοιχείο. Θα ήταν ίσω σκόπιμο οι νομοθέτες να εξετάσουν αν κανονισμοί ακριβώς ε, μεταξύ αυτών των δύο σωμάτων θα πρέπει να συνεξετάζονται σε μια συνάρτηση, σε μια αλληλεξάρτηση. Επιπλέον πρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις που έχουμε με την όλα την ομάδα τον Οργανισμό Καταπολέμησης Απατών ως κύριο εταίρο για την καταπολέμηση των απατών ακριβώς ε, κατά τον ε, εις βάρος των συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γίνει δουλειά εκεί για να βελτιωθούν τα πράγματα και σίγουρα ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν να βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια στο μέλλον. Επιπλέον έχουμε συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη να οικοδομήσουμε σε, πάνω στις σχέσεις που ήδη έχουμε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την COSIC, ε, την ε, Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια. Η Eurojust συνεισφέρει με σοβαρό τρόπο στις διαβουλεύσεις ε, και δράσεις της COSIC υπό το άρθρο 71 ακριβώς της συνθήκης της Λισαβόνας. Και θα έλεγα ότι είναι σημαντικό, όπως πιστεύω, να υπάρχει μια δικαστική συνεισφορά στις διαβουλεύσεις της ΚΟΣΙΚ υπό ένα πρίσμα τουλάχιστον φαίνεται να ακολουθεί την συνιστόσα την παράμετρο της επιβολής του νόμου στις διαβουλεύσεις της. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η δικαστική παράμετρος. Μία πτυχή λοιπόν αυτής της εταιρικής σχέσης όπου η Eurojust θα έλεγα μπορεί να δράσει σωστά είναι ως ένας κεντρικός εταίρος, αν όχι ο κεντρικός εταίρος, ο κύριος εταίρος στην καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτός ο τομέας είναι ο τομέας των ομάδων κοινών ερευνών, joint investigation teams. Ε, είμαστε τώρα μέλος ε, της γραμματείας για, αυτές, ε, για αυτούς τους αξιωματούχους επαΐοντες των κοινών ομάδων ερευνών διακρύβωσης. Επίσης παρέχουμε και κονδύλια, επικουρούμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες ερευνών. Επίσης όσον αφορά και κονδύλια της Ευρωπαϊκής που με βάση την πραγματογνωμοσύνη και πείρα που έχουμε συλλέξει στη Eurojust για το πού θα μπορούσαν με τον καλύτερο τρόπο να κατανεμηθούν αυτά τα κονδύλια όσον αφορά τις κοινέ ομάδες ερευνών όλα αυτά ήταν μια επιτυχία, επιτυχής πρωτοβουλία. Στην ετήσια έκθεσή μας θα δείτε ότι η Eurojust συμμετείχε σε 20 περίπου τόσες ομάδες ερευνών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 2010. Επίσης υποστηρίζουμε πόσες περίπου, 25, 22 θα έλεγα, κοινέ τέτοιε ομάδες ερευνών και διακρύβωσης που προσήλθαν στην Eurojust με αιτήματα χρηματοοικονομικής ε, υποστήριξης. Δεν είναι μόνο τα κονδύλια που τους δίνουμε, τους δίνουμε και πραγματογνωμοσύνη της γνώσης μας, ώστε να υπάρξουν με σωστό τρόπο οι συμφωνίες για αυτές τις κοινέ ομάδες ερευνών και να υπάρχει αποτελεσματικό, θετικό αποτέλεσμα στην καθημερινή προσπάθεια προσπάθεια καταπολέμησης του διοργανωμένου, του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Σε αυτά νομίζω ίσως μακρηγόρησα και ξεπέρασα το χρόνο μου. Ζητώ συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Φοβερή παρουσίαση αυτή που ακούσαμε. Και τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση. Από ό,τι κατάλαβα, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόντες, αλλά δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε αυτή τη φάση της συζήτηση. Οπότε, η κυρία Βέμπερ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Άλετ Βίλιαμς για την παρουσίασή του. Είναι γεγονός ότι έπρεπε να μας υπενθυμίσει κάποιος ε, την εργασία της ε, Eurojust ε, και σε σχέση με τη δραστηριότητά σας θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι αυξήθηκαν και οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολείστε αλλά αυξήθηκαν και τα αποτελέσματα τα καλά αποτελέσματα των εργασιών σας. Ε, εκτιμώ το γεγονός ότι θέλετε να νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο συνεκτικό τρόπο και εγώ αυτό θα ήθελα για το μέλλον. Αλλά αν με ρωτήσετε πόσο αισιόδοξη είμαι, θα έλεγα ότι από αυτά που έχω δει τα τελευταία χρόνια δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη. Οπότε δεν μπορώ να πω αν για παράδειγμα η ανεθεώρηση, η μεταρρύθμιση της ε, Eurojust και της ε, Europol ε, θα συνάδουν, ελπίζω τουλάχιστον να υπάρξει μια συνοχή. Έχω δύο ερωτήσεις γιατί θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα. Όταν αναφερθήκατε βέβαια στην προστιθέμενη αξία γενικότερα της συνεισφοράς της Eurojust, δεν προσπαθώ να οδηγήσω τη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όταν μιλάμε για οικονομικό έγκλημα. Έχουμε ας πούμε μια χώρα, η Δανία, που έχει επαναφέρει τους εσωτερικούς ελέγχους, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του διασυνοριακού εγκλήματος. Έχετε ε, την εντολή να ασχοληθείτε με τέτοιου είδους υποθέσεις. Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό αυτή η επαναφορά των εσωτερικών ελέγχων είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Επίσης αναφέρθηκατε ε, στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Καταλαβαίνω βεβαίως ε, το βαθμό στον οποίο θεωρείτε εσείς ότι, ήταν, ε, είναι σημαντικό αυτό. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποιους δισταγμούς σε σχέση με το πόσο αποτελεσματικό ήταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως τώρα. Γιατί υπάρχουν πολλέ, πολλοί ισχυρισμοί καταχρήσεων, ειδικότερα όταν μιλούμε για την αρχή της αναλογικότητας και τη διατήρησή της. Χθε ακούσαμε, ας πούμε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, της Πολωνίας, που ήταν εδώ, και όταν τον ρωτήσαμε ειδικότερα για την αναλογικότητα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Οτιδήποτε είναι πάνω ε, ε, από, ε, σημαίνει πάνω από ένα χρόνο φυλάκιση, μπορεί να είναι αντικείμενο ευρωπαϊκού εντάλματο συλλήψεω. Η, η άποψή μου λοιπόν, και υποθέτω ότι αρκετοί συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου, ότι έχουμε ίσω διαφορετική κατανόηση τη αναλογικότητα. Τι, τι είναι σοβαρό αδίκημα και αν το σοβαρό αυτό αδίκημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα δικαιοδοσίας, αλλά θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Όσον αφορά τώρα τις ε, κοινέ ομάδες, τις ερευνητικές, ε, καταλαβαίνω ότι είναι ένας ε, χρήσιμος μηχανισμός, αλλά το ερώτημά μου έχει να κάνει με την προστιθέμενη αξία σε σχέση με το χρόνο. Πόσο χρόνο εξοικονομείται όταν συμμετέχει στην όλη διαδικασία ε, όταν συμμετέχει στην όλη διαδικασία Eurojust. Και ελπίζω ότι κάποια αντιπροσωπεία από εμά θα έρθει στη Eurojust να συζητήσει περισσότερο το θέμα αυτό με εσά για τους συναδέλφους σας. Η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίλιαμς. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας και πραγματικά με μεγάλη προσοχή θα διαβάσω την έκθεσή σας. Δεν τα άκουσα βέβαια όλα όσα είπατε γιατί ήρθατε λίγο νωρίτερα και εγώ καθυστέρησα. Νομίζω ότι στους στρατηγικούς σας στόχους και στα στρατηγικά σας ε, σχέδια, στο σχετικό έγγραφο αναφέρετε ότι θέλετε να συνεχίσετε τη βελτίωση της συνεργασίας μέσω ενεργού ε, Υποβολή ε, συστάσεων ε, στους υπεύθυνου λήψη αποφάσεων στην, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα ήταν πολύ χρήσιμο και για μα αν έρχονται οι διάφοροι φορείς να μας εξηγούν τι ακριβώς κάνουν και όταν έχουν και συγκεκριμένες ιδέες για βελτίωση. Αλλά πώς μπορείτε να είστε τόσο δραστήριοι όσον αφορά τα ζητήματα ε, του Ευρωπαίου Δημοσίου Κατηγόρου, γιατί αναφέρετε ότι ήταν πάρα πολύ σημα... είναι πολύ σημαντική η ενεργό συμμετοχή της Eurojust βάσει του άρθρου 6 κλπ. κλπ. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι ακόμη πεπισμένη σε σχέση με αυτό. Με τη χρησιμότητα, εν πάση περιπτώσει, ε, της ε, ιδιότητας αυτής και θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Ε, και όπως είπε και η κυρία Βέμπερ, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που, που, κάνατε για το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης, θα ήθελα να μας πείτε σε σχέση με την εμπειρία που είχατε αν θεωρείτε κατά πόσο είναι ζήτημα ε, δημοσίου συμφέροντος μερικές φορές να αποφασιστεί αν κάποιος ε, θα κατηγορηθεί μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως ή όχι και ότι και πώς ε, συνεισφέρει η Eurojust σε αυτήν την διατήρηση της αναλογικότητας Εσείς βασίζεστε στις αξιολογήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου σε σχέση με το πόσο καλά λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη. Θα θέλαμε να μας πείτε σε σχέση με την Europol ποιο είναι το πρόβλημα με την επιχειρησιακή συνεργασία. Δεν θυμάμαι ακριβώ πώς το είπατε, αλλά μου φαίνεται ότι η, από ό,τι μας είπατε τουλάχιστον έχει κάποιες επιφυλάξεις η Europol και σας μεταχειρίζεται ως ε, τρίτο ε, στην προτεραιότητα εταίρο. Οπότε δεν ξέρω Μήπως θα έπρεπε κάπως να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο της ε, συνεργασίας αυτής. Αυτά ήθελα να ρωτήσω σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα κάτι να προσθέσω και για το ένταλμα συλλήψεως. Εντάξει, είμαι υπέρ σε γενικές γραμμές, αλλά ως Ευρωβουλευτής που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, και γνωρίζετε ότι έχω πολλές φορές ακούσει διάφορες περιπτώσεις ε, υποθέσεων που είναι ε, ε, νομικώς πολύ επίμαχες και όταν ε, γνωρίζουμε κιόλας κάποιον άνθρωπο, για παράδειγμα ένας συμπολίτης μου από το Λονδίνο τελικά θωώθηκε στην Ελλάδα, Εν πάση περιπτώσει <coughs> ήταν μια τεράστια περιπέτεια αυτή από την οποία πέρασε, θα το γνωρίζετε και ίσως θα μπορούσατε κι εσείς να μας πείτε τη δική σας εμπειρία, γιατί είναι γεγονός ότι η αμοιβαία αναγνώριση των ε, δικαστικών αποφάσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, δεν ήταν επαρκής για τη βελτίωση ε, ε, των ε, της ποινική δικαιοσύνης και τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση με τα ε, δικαιώματα ε, του κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας. Τι νόημα λοιπόν έχει να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους αλλαγές αν δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αν δεν χρήζει ευρείας αποδοχής από το κοινό. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στους επένους και την εκτίμηση προς τον πρόεδρο της Eurojust, κύριο Williams, για δύο απλούς λόγους. Η έκθεση είναι πραγματικά πολύ πλούσια, πολύ ενδιαφέρουσα και η σύνθεση είναι πολύ πετυχημένη και ωραία διευκολύνει και τους δικούς μας προσανατολισμούς και τη δική μας αναζήτηση με τα διάφορα κεφάλαια και κατηγορίες. Και υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Η ερμηνεία του Προέδρου καμιά φορά είναι πιο ενδιαφέρουσα από το συστατικό τμήμα πολλών στοιχείων όσον αφορά και τα στατιστικά. Στατιστικά. Είδα ένα κατάλογο στη σελίδα 29. Τι λέει, τι δείχνει. Καταδεικνύει τις περιπτώσεις. Τον αριθμό των περιπτώσεων δίμευσης και κατάσχεσης όσον αφορά κονδύλια, χρήματα τα οποία κατασχέθηκαν ή δημεύθηκαν το 2010 ο κατάλογος, ο πίνακας είναι πίνακας κάποιων περιπτώσεων. Αυτές οι περιπτώσεις είναι η ερώτησή μου, είναι οι πιο σημαντικές, οι πιο οι ευρύτερες όσον αφορά την ετήσια δραστηριότητά σας ως θεσμικού οργάνου της Eurojust. Αν όχι, είναι δυνατόν στην επόμενη ετήσια έκθεση να μας δώσετε έναν πιο επεξηγηματικό, πληρέστερο, πιο εξαντλητικό πίνακα με τις περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει όλες να συμπεριληφθούν και να δημοσιευθούν για να είναι στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Και δεύτερον, κατανοούμε ότι σε σχέση με την δίμευση ή κατάσχεση χωρίς καταδίκη είναι ένα πολύ επίμαχο σημείο, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Και συνδέεται όχι μόνο απλά με παραδοσιακούς περιορισμούς όσον αφορά την ομοθεσία ή τα συντάγματα αυτών των κρατών μελών, αλλά το επίμαχο θέμα για αυτό το μηχανισμό, για αυτές τις διεργασίες ή διαδικασίες δικονομικά είναι αποτέλεσμα σε σχέση με την ε, λιγότερη ε, ανάπτυξη, μικρότερη ας το πούμε έτσι ε, εκλέπτυνση ή ανάπτυξη διότι το πάγωμα ή κατάσχεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων σημαίνει πολλές φορές την καταδίκη και την χρεοκοπία πολλών τέτοιων ανθρώπων. Αυτό με βάση την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, χωρίς δηλαδή να υπάρχει καταδίκη δικαστική, δεν μπορεί να γίνεται. Στην επόμενη σελίδα διαβάζουμε ότι το 2010 η Eurojust ε, εξέτασε τέτοιου, με, τέτοιου είδους χωρίς ε, νομική ε, καταδίκη, κατάσχεση ή δίμευση ως αμφισβητήσιμη. Μετά έχουμε κράτη-μέλη τα οποία δεν τοποθετήθηκαν λέει και δεν απήντησαν και τους πιθανούς ε, λόγους για την απουσία απαντήσεων και τοποθέτησης από πλευρά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένετ παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ για την, για την παρουσίασή σας. Ήταν αναλυτική και μας βοηθάει να εκτιμήσουμε μια δουλειά που δεν την αναγνωρίζουμε λόγω άγνοιας τελικά. Μου τράβηξε ιδιαίτερα την ε, προσοχή όταν ε, μιλήσατε για, ε, για την τηλεφωνική παρακολούθηση. Πολύ συχνά ρωτιούνται τα κράτη-μέλη σχετικά από τα μέσα μαζική. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μία μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκλοπές ως απόδειξη. Θέλω να ξέρω πόσο σημαντικές είναι στην ανταλλαγή δεδομένων και πώς οι υποκλοπές μπορούν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τι κάνετε για την καταπολέμηση της ε, κυβερνοεγκληματικότητας και πώς μπορείτε να παλέψετε ουσιαστικά κατά της τρομοκρατίας και ποιο ρόλο θα μπορούσατε να αναλάβετε πιο βασικά δηλαδή για την καταπολέμηση αυτής της απειλής στην Ευρώπη. Δεν βλέπω άλλους ε, που να θέλουν το λόγο. Ο πρόεδρος της Οπότε δίνουμε και πάρει το λόγο στον κύριο σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα ευγενή σχόλια, τα ευγενή και ευνοϊκά σχόλια και τα, τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω <clears throat> τα σχόλια με κάποια συγκεκριμένη σειρά ανάλογα με τις σημειώσεις μου. Ζητώ συγγνώμη αν δεν καλύψω όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις σας. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα της κυρίας Βέμπερ, το πρώτο θέμα σε σχέση με την αποκατάσταση των συνοριακών ελέγχων, θα προσπαθούσα να αποφύγω, ζητώ κατανόηση άμεσα αυτή την, απάντη, την ερώτηση που έχει τόσο, τόσες πολλές ε, πολιτικές επιπτώσεις ε, και μεγάλη πολιτική σημασία. Τώρα, όσο αφορά τη Eurojust, το σκεπτικό για τη Eurojustice ήταν να παράσχει μια αντισταθμιστική δράση η εξισορρόπηση για την ε, ελευθερία κυκλοφορίας όσον αφορά <laughs> τους εγκληματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ε, συνέπεια της ε, κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η δράση της Eurojust. Υπάρχει για να ελέγχει και να δρά ώστε οι διοκτικές αρχές και οι ερευνητικές αρχές να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε κάποιο βαθμό, α το πω έτσι, ώστε άμεσα να μπορούν να αντιδράσουν και να δράσουν και εξίσου ταχαίως να μπορούν άμεσα ταχύτατα να δράσουν δράσεων, διώκοντας, καταδιώκοντας τους ε, εγκληματίες. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο σε κάποιο βαθμό και αυτό απηχήθηκε στα σχόλια της Βαρονέσας Λαντφόντ. Σαφώς υπάρχει ένα θέμα εδώ όσον αφορά την αναλογικότητα. Και αυτό είναι κάτι που τακτά και σε τακτό επίπεδο θίγεται και αναφέρεται. Στις περιπτώσεις της Eurojust τώρα, πρέπει εδώ να ομολογήσω και να πω ότι αυστηρά υπό τους όρους του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης πρέπει σαφώς να αντιμετωπίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπως υφίσταται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεταθέσεις ή μεταφορές που έχουν υπάρξει στα κράτη-μέλη νομοθετικά, νομικά. Το θέμα της αναλογικότητας δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο απόφασης για το ευρωπαϊκό ένταλμα θα μπορούσε κανείς λογικά να επιχειρήσει και να πει υπό το άρθρο 49 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί η αναλογικότητα σύμφωνη εντάξει αλλά δεν είναι κάτι επί του οποίου Eurojust είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ξεχωριστά πέρα από το να διασφαλίσει ότι τα επιχειρήματα αμφωτέρωθεν θα πρέπει να είναι γνωστά και να ε, με βάση αυτά να προχωρούμε. Αυτό που συνέβη είναι με βάση την πείρα και την εμπειρία εμπειρία της Eurojust, αυτά που συλλέξαμε ως στοιχεία και συμπεριλαμβάνονται στα τεκμήρια, στα στοιχεία τα οποία έχουν διαβιβάζονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εγχειρίδιο για παράδειγμα, το οποίο συνοδεύει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Εξίσου λοιπόν σημαντικό για το μέλλον αυτό το στοιχείο, για αυτή τη δουλειά και για τις συζητήσεις που αφορούν τις, ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερευνών ή ανακριτικών ερευνών. Και τώρα με επίκεντρο τις δυσκολίες που διαγνώσαμε όσον αφορά τη δυσκολία για την αναλογικότητα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Τώρα λοιπόν θα υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση και διάταξη από ό,τι γνωρίζω ανάλογα με την τελική νομοθετική απόφαση που θα ληφθεί και θα, θα απαιτεί αυτό από τα κράτη-μέλη να εκδίδουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα ότι θέματα αναλογικότητας νομοθετικά ή νομολογικά έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν αντιμετωπιστεί. Και η Eurojust έχει παράσχει εκείνο το οποίο πιστεύω ότι είναι μια θετική συνεισφορά για τη συζήτηση, για τη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Ερευνών και το θέμα της αναλογικότητας που καλύπτει αυτό το ζήτημα, πρέπει να καλύπτει. Τώρα όσον αφορά το θέμα που ε, αφορά τις κοινέ ομάδες ε, ερευνών η πείρα της Eurojust θα έλεγα είναι ότι είμαστε σε θέση από το γεγονός της ίδιας της διάρθρωσης και δομής δημιουργίας αυτών των ομάδων καταφέραμε να επιβραχύνουμε, να ε, μειώσουμε το χρονικό ε, διάστημα από την ε, συγκρότηση μέχρι την λειτουργικότητα αυτών των δράσεων. Ένα από τα στοιχεία είναι ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα στην ομάδα θα είναι διαθέσιμα σε όλη την ομάδα. Δεν θα είναι πλέον αναγκαίο υπό το πλαίσιο μιας κοινή ομάδας ερευνών να εκδίδονται αιτήματα ξεχωριστά τα οποία θα εγκρίνονται στη συνέχεια και όπως σωστά αναφέρθηκε αυτό ήταν ένα, ένας από τους κύριους λόγους καθυστερήσεων για την απόκτηση τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων διασυνοριακά. Όλα τα προβλήματα που είχαν σχέση με τον, τη σύνταξη, την ε, μετάφραση, την διαβίβαση αυτών των αιτημάτων οδηγούσαν σε καθυστερήσεις και όλα αυτά τώρα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν με την άμεση δράση των κοινών ομάδων ερευνών. Η Eurojust ακριβώς ως επίκεντρο της πραγματογνωμοσύνης για αυτές τις κοινέ ομάδες ερευνών θα διασφαλίσει ότι αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι μια θετική συνεισφορά θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά της. Αυτά για τα σημεία που αφορούν τον συσχετισμό <clears throat> με τις ε, ευρωπαϊκές διοκτικές αρχές τώρα για την εισαγγελία. Η Eurojust δεν έχει μια θέση που θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς λέγοντας ναι ή όχι, υπέρ ή κατά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και νομίζω ότι θα έλεγα ότι δεν είναι συνήθιστο αυτό. Είμαστε ένα σώμα πρακτικό πρακτικής υλοποίησης και εφαρμογής που ασχολείται με τέτοιου είδους περιπτώσεις. Έργο αυτής της φύσης ε, υπέρ ή κατά αυτό, αυτής της αρμοδιότητας θα πρέπει να επιλύεται από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως π.χ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Eurojust είναι να εξετάσει τις περιπτώσεις της και να ταυτοποιήσει να εντοπίσει προβλήματα τα οποία εμπειρικά διαπιστώνουμε ότι υφίστανται όσον αφορά για παράδειγμα την ε, ε, υπονόμευση οικονομικών συμφερών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούμε στο μέλλον να μπορέσουμε με τα συμπεράσματα που συνάγουμε να τα διαθέσουμε στους νομοθέτες ώστε να αποφασίσουν εκείνοι για το τι πρέπει να γίνει για τέτοιες περιπτώσεις. Εξίσου αφορώντας το στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε, την παρέμβαση που έγινε όσον αφορά το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και της ανάγκης να διασφαλίσουμε κατά κάποιο τρόπο ότι θα υπάρχει και εμπιστοσύνη αλλά και σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ελπίζω να μην παρεμήνευσα την παρατήρησή σας, κυρία ή κύριε, αυτή την παρατήρηση που κάνατε εσείς. Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της συμμετόζει η Eurojust θέλει με κάθε τρόπο να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει η δικαστική παράμετρος λήψης υπόψη δικαστικών θεμάτων και δικαιωμάτων όσον αφορά την ε, στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω πραγματικά είμαστε το μόνο όργανο το οποίο μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και να διασφαλίσει αυτή την πτυχή αυτών των δικαιωμάτων και δικαστικών παραμέτρων. Και εξίσου παράλληλα παράλληλα έχουμε προαγάγει και υποστηρίξει έναν φορέα, ένα σώμα που πρόσφατα συγκροτήθηκε. Το Συμβουλευτικό Φόρουμ, το Συμβουλευτικό Βήμα των Γενικών Εισαγγελέων και Διοκτικών Αρχών. Εκεί συγκλίνουν και συνέρχονται οι επικεφαλείς όλων των διοκτικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζονται μεταξύ τους. Μέσω της ε, εταιρική ε, σχέσης είναι μέλος η Eurojust στην Κόζη και υπό το άρθρο 71 η συμμετοχή μας σε τέτοιου είδου τους ε, εγχειρήματα για την εσωτερική ασφάλεια, στην εσωτερική αρχιτεκτονική, μέσα στο σώμα αυτών ακριβώς των επικεφαλής διοκτικών αρχών και εισαγγελιών, με το μέλημα να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτά τα στοιχεία να είναι σεβαστά. Η παρέμβαση, η παρατήρηση που έγινε σε σχέση με το συσχετισμό μας με την Ευρωπόλ, τη Europol ως Eurojust, Θέλω να πω ότι καθώς δεν εκφράστηκα ίσως με τη σαφήνεια που θα έπρεπε να είχα υιοθετήσει η θέση μας όσον αφορά τη Eurojust σε σχέση με την Ευρωπόλ λειτουργούμε σε ένα λειτουργικό επίπεδο, έτσι δρούμε. Αλλά θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα θεσμικά προσκόμματα ή εμπόδια που μπορούν να αφαιρεθούν, να αρθούν ακόμα στο μέλλον. Και αναλύοντας ε, τις περιπτώσεις όσον αφορά το συσχετισμό μας, τη σχέση με την Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ συλλέγει όπως γνωρίζετε στοιχεία δεδομένα από τα κράτη-μέλη και κατηγορίες ή ομάδες αυτών των στοιχείων ή δεδομένων ανάλογα με κατηγορίες εγκληματικών περιπτώσεων. Παράδειγμα, εμπόριο ανθρώπων, παράδειγμα, λαθρεμπόριο, προϊόντα απομίμησης, μαϊμούδε εκμετάλλευση ανθρώπων, εμπορία ανθρώπων και τα λοιπά συναφή. Και <clears throat> ενώ υπάρχουν προτάσεις να υπάρξει μια μετάθεση περίπου 22 τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια αναλύσεων ε, σε, ε, από αυτά η, η Europol ε, με 15 από αυτές τις αναλύσεις εμπλέκεται και θα ελπίζαμε αν θα υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο επανεξέτασης του καθεστώτος μας αυτό θα ήταν αυτόματα να γινόμαστε άμεσα συνδεδεμένοι και άμεσα να συνδεόμαστε με το, την ανάλυση αυτού του έργου από πλευράς της Ευρωπόλ. Είναι θέμα ε, τοποθέτησης και βούλησης όσον αφορά την ε, Ευρωπόλ. Πρέπει να το δούμε. Θα μπορούσε ε, να υπάρξει αυτή η σύνδεση και η εταιρική σχέση. Αυτό φυσικά πολλές φορές εξαρτάται και από αποφάσεις των κρατών μελών. Και γι' αυτό έθεσα την ιδέα, πρότεινα την ιδέα να εξεταζόταν μια ρύθμιση ώστε να μπορούσε από πλευράς Ευρωπόλ να θεωρηθεί αυτονόητη μια τέτοια εταιρική σχέση, μια τέτοια σύνδεση. Τώρα, όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρατε εσείς για τη σελίδα 29 της έκθεσής μας, για αυτόν τον κατάλογο, αυτός ο κατάλογος είναι μια περίληψη, επιλεκτικός κατάλογος περιπτώσεων ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται με αυτή τη μορφή και τρόπο είναι ότι η έκθεσή μας πάντα συντάσσεται έχοντας υπόψη το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε να, να δώσουμε στοιχεία για περιπτώσεις που βρίσκονται υπό εξέταση από πλευράς μας. Δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ή δημοσιοποιήσουμε τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν τέτοιες ε, πιο σημαντικές περιπτώσεις αλλά δεν έχουμε την ελευθερία να τις ε, εγγράψουμε, να τις ε, δημοσιοποιήσουμε στην ετήσια έκθεσή μας. Ίσως στο μέλλον θα είναι δυνατόν να έχουμε και περισσότερα παραδείγματα που θα σας δίνουμε. Τώρα, το σημείο να μην υπάρχει κατάσχεση ή δίμευση χωρίς νομική καταδίκη από δικαστήριο είναι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την έκθεση και κατανοώ ότι θέτει και δημιουργεί πολύ σημαντικά ζητήματα, ζητήματα αρχής, επιθεμάτων αρχής. Η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν μια προσέγγιση χωρίς ε, ε, να απαιτείται η νομική καταδίκη, η δικαστική καταδίκη για δίμευση ή κατάσχεση. Μπορούν και τη ερήμην ε, του κατηγορούμενου και σε σχέση με τις, την δίωξη να κατασχεθούν ή να δημευθούν. Αυτό δημιουργεί θέματα όπως αναφέρθηκε όσον αφορά το τεκμήριο της αθωότητας που υφίσταται πάντα δικαστικά. Υπάρχουν επιχειρήματα για το τεκμήριο το άρθρο 6 για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν θίγεται από αυτού του είδους ε, της ε, ε, κατασχέσης ή δημεύσης χωρίς δικαστική καταδίκη. Και εδώ απλά σχηματικά και συνοπτικά μπορώ να αναφέρω το εξή. Ένα επιχείρημα. Η δίμευση τέτοιων ε, προϊόντων ή τέτοιων περιουσιακών στοιχείων <clears throat> δεν είναι κάτι το οποίο συνεπάγεται, ε, ε, γίνεται με βάση την αθωότητα ή όχι. Γίνεται απλά δράση εις βάρος περιουσιακών στοιχείων ενός ατόμου. Και έτσι το τεκμήριο της αθωότητας εδώ δεν έχει άμεση εφαρμογή και ένα άλλο ε, επιχείρημα είναι ότι δικονομικά στα κράτη-μέλη, στα τέσσερα αυτά κράτη-μέλη που έχει, ε, ισχύει για αυτά η μη καταδίκη, ως δηλαδή η ε, δίμευση μπορεί να προχωρήσει χωρίς καταδίκη, είναι αστικού χαρακτήρα και όχι ποινικού χαρακτήρα. Σε σχέση δηλαδή με την ε, προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και την αρχή αυτή δεν θα εφαρμοστεί και σε σχέση με την τελευταία παρέμβαση που έγινε από την ε, Ευρωβουλευτήνα, από την Ισπανία, το ερώτημα σε σχέση με τις ε, συλλογές στοιχείων ε, και παρακολουθήσεις και την καταπολέμηση τρομοκρατικών δράσεων από πλευράς Eurojust έχουμε μια πολύ δραστήρια ομάδα καταπολέμησης ε, των τρομοκρατών και της τρομοκρατίας στην Eurojust. Πέρυσι είχαμε θα έλεγα νομίζω πέντε συντονιστικές συνεδριάσεις όπου είχαμε απεσταλμένους πραγματογνώμενες από τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένες περιπτώσεις για να προαχθεί στο επίπεδό μας η καταπολέμηση των, τρομο τρομοκρατών. Έχουμε όμω και στρατηγική ε, σημασία τέτοιε συναντήσει. Κάθε κράτο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται να έχει ένα σύνδεσμο σε εθνικό επίπεδο που θα έχει καθοριστεί σε σχέση με το έργο τη Eurojust. Ελπίζουμε αυτή η συνάντηση στη Χάγη στην Ολλανδία να ε, φέρει την πραγματογνωμοσύνη των εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη ώστε να εργαστούμε με τον πιο θετικό τρόπο. Και έτσι σε συγκεκριμένα θεματικά προβλήματα θεματολογικά θα επικεντρωθούμε όσον αφορά για παράδειγμα την δράση και των ε, ε, τρομοκρατών ε, και όσον αφορά την κυβερνοτρομοκρατία παρότι εξετάζουμε αυτό το θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ακόμα να περαιτέρω να αναπτυχθεί στην Eurojust. Οι κυβερνοτρομοκρατικές δράσεις είναι κάτι που είναι δύσκολο ίσως να μετρηθούν υπό στατιστικό πρίσμα κάποιοι οι οποίοι ε, άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονται κάποιοι ή κάποιοι που ε, μπορούν να, στο διαδίκτυο να ακολουθούν κάποιους τρομοκρατικούς στόχους μπορούν να καταχωρούνται ίσως στατιστικά σε διαφορετική κατηγορία σε σχέση με το κυβερνοέγκλημα. Έχουμε στοιχεία, δεν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και αυτό ειλικρινά ομολογώ επειδή πολλές φορές ε, έχουμε, όταν έχουμε περιπτώσεις τρομοκρατικών δράσεων έχουμε διαφορετικές κατηγορίες ε, καταχώρησης ε, και όχι υποχρεωτικά την κατηγορία στατιστικά των εγκλημάτων. Ελπίζω να απάντησα. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Williams. Ήταν πραγματικά μια διεξοδική παρουσίαση. Σα συγχαίρω, δεν σας επιπλήττω. Πραγματικά ήταν πολύ καλή η παρουσίασή σας, της ε, ετήσιας έκθεσή σας. Ήταν μια πολύ ε, χρήσιμη και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ε, ελπίζουμε να ε, μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τη συνεργασία μας και στο μέλλον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ασφάλειας, Δικαιοσύνης και Ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα περιμένουμε εναγωνίως την ε, επόμενη συνάντησή μας ε, μαζί σας. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Φρανσουάζ Λεμπάι, εκ μέρους